Uh, good afternoon. Καλό σας απόγευμα, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Εδώ έχουμε επίσης web streaming ε, όσον αφορά την ε, συγκεκριμένη μας ε, συνεδρίαση. Γι' αυτό λοιπόν δεν θέλουμε να αργοπορήσουμε και πολύ. Πρέπει να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Ήδη είναι 3 και 10 και επομένως πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσουμε την συνεδρίασή μας. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω ότι έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα σημεία στη μέση διάταξή μας. Για την επόμενη μία ώρα λοιπόν θα έχουμε τη χαρά θα έχουμε τη χαρά λέω να συναντήσουμε την ε, Λουξεμβουργιανή Προεδρία μέσω του κυρίου Μάρκ Χάνσεν του Υπουργού που είναι υπεύθυνο για θέματα έρευνας. Πρέπει να σας πω κύριε Υπουργέ ότι το πρωί είχαμε τον Πρωθυπουργό σας εδώ στην ε, αίθουσά μας και μάλιστα ε, τώρα είναι ακόμα μεγαλύτερη η χαρά μας που συνεχίζονται οι ε, οι επισκέψεις ε, από πλευράς του Λουξεμβούργου. Θα μας μιλήσετε για θέματα καινοτομίας και έρευνας. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά για μας. Και στην Επιτροπή μας, στην Επιτροπή Ήτρε λοιπόν, αισθανόμαστε υπεύθυνοι για το θέμα αυτό και επομένως συνεργαζόμαστε στενά με την Επιτροπή ε, για θέματα έρευνας και ε, τεχνολογίας και θα θέλαμε τώρα να ακούσουμε τις προτεραιότητές σας στη διάρκεια του εξαμήνου της Προεδρίας σας. Παρακαλώ λοιπόν να πάρετε το λόγο και να μας κάνετε την αρχική σας παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής κυρίες και κύριοι. Νομίζω πως όλοι γνωρίζετε ότι την 1η Ιουλίου ανέλαβε τα Ινία της Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για 12η φορά, ε, για η φορά ε, το Λουξεμβούργο. Ε, εγώ θα ήθελα να παρουσιάσω το πρόγραμμα έρευνας και επιστήμης ε, το οποίο έχουμε σχεδιάσει ε, με τρόπο ώστε να απελευθερώσει δυνάμεις και δυναμισμό για το δεύτερο εξάμεινο του τρέχοντος έτους. Εμείς θέλουμε σωστή διακυβέρνηση, ισότητα ανδρών γυναικών στην έρευνα ε, και ακαιρεότητα της έρευνας. Πριν ε, περάσω στην ουσία του θέματος, θα ήθελα εν συντομία να σας παρουσιάσω το Εθνικό Σύστημα Ερεύνης στο Λουξεμβούργο. Έχουμε τρία μεγάλα δημόσια ερευνητικά κέντρα, τα οποία δημιουργήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 80 έχουμε ένα πανεπιστήμιο, ε, το οποίο υπάρχει εδώ και 12 χρόνια μόνο και ε, το κράτος δίνει 315 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ε, να σας πω ας πούμε ότι το 2000 μονάχα 27 εκατομμύρια έδινε ε, το κράτος για τα ερευνητικά κέντρα και το πανεπιστήμιο. Έχουμε αυτοί 200 ερευνητές που δουλεύουν στο Λουξεμβούργο. Τον δε ε, Σεπτέμβριο με περηφάνεια ε, θα εγγενιάσουμε την ε, το κάμπος του Μπέλβαλ ε, για το οποίο είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι και το οποίο θα αποτελέσει κοιτίδα έρευνας καινοτόμων ε, επιχειρήσεων και εταιριών και είμαι πάρα πολύ περήφανος γιατί θα αποτελέσει και στα σταυροδρόμι των δημοσίων και ιδιωτικών ερευνών. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας είναι ιδιαίτερος προσφυλής στο Λουξεμβούργο. Επανειλημμένα ζητήσαμε σε διάρκεια συμβουλίων την ολοκλήρωση αυτού του χώρου. Ε, εμείς θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε ε, στην διαδικασία αυτή ε, αυξάνοντας τον συντονισμό και τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, θεωρούμε ότι η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη ε, πρέπει να συμβάλλουν ε, σε εταιρική σχέση στην ανάπτυξη αυτού του χώρου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρουσιάσει δύο εγγραφά όσον αφορά τον ε, ερευνητικό ε, ενιαίο χώρο ε, και πρέπει να σας πω ότι η έρευνα και η καινοτομία δυστυχώς είναι χώροι που ακόμα είναι κατακαιρματισμένοι και επομένως δεν δίνουν την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εκμεταλλευτεί τα αποτελέσματα της Ένωσης της Έρευνας σε συνεργασία με την Κομισιόν και με την ε, βοήθεια του Βεράκ ε, στους 18 τελευταίους μήνες έχει δημιουργηθεί, έχει εκπονηθεί ε, ο οδικός χάρτης μέχρι το 2020. Πρόκειται για οδικό χάρτη ο οποίος εγκρίθηκε η Πολετονική Προεδρία στις 29 Μαΐου τρέχοντος έτους και περιλαμβάνει μέτρα τα οποία μπορούν θετικά να έχουν επίπτωση στην έρευνα και επομένως να ε, ε, συμβάλλουν θετικά στη δημιουργία του ευρωπαϊκού χώρου τα κράτη-μέλη καλούνται μέχρι το 2016 να ε, ε, εγκρίνουν τους εθνικούς οδικούς χάρτες και να καταρτήσουν κατάλογο ε, συγκεκριμένων δικτών από κοινού με το ΕΡΑΚ έτσι ώστε να έχουμε την δυνατότητα να μετρήσουμε τις πρόοδους σε συγκεκριμένους τομείς. Πριν αναφερθώ στην, ε, στο ίδιο το θέμα, επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επανέλθω στην προτεραιότητα 4 του οδικού χάρτη, δηλαδή η ισότητα φύλων και ε, την ε, ε, ισομερή συμβολή ανδρών και γυναικών στην έρευνα. Αυτό θα είναι ένα από τα δύο θέματα που θα συζητήσουν οι αρμόδιοι υπουργοί στην άτυπη συνεδρίαση την επόμενη Τρίτη στο Λουξεμβούργο, της οποίας θα έχω την χαρά και το προνόμιο να προεδρεύω. Σήμερα το πρωί έμαθα ότι η Επιτροπή Δικαιωμάτων της Γυναίκας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε χθε μια έκθεση ε, σχετικά με την ανάγκη να ξεπεράσουν ε, οι γυναίκες αυτά τα αόρατα εμπόδια ε, που τους φράσουν την πρόσβαση στην επαγγελματική τους ζωή. Επομένως καταλαβαίνω ότι είναι πολύ επίκαιρο το θέμα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα δεύτερο σημείο επίκαιρο, το οποίο θα ήθελα να υπογραμμίσω, ε, είναι ένα ε, άρθρο το ε, γερμανικό περιοδικό Der Spiegel ε, στην έκδοση αυτής της εβδομάδας ε, αναφέρεται στην κυρία, στις κυρίες Μόζερ και Φόλερ οι οποίες πήραν το βραβείο Νόμπελ και που συζητούν και αναφέρονται στην ισότητα των ανδρών και γυναικών και που λένε ότι ακόμα δρόμος υπάρχει που πρέπει να γίνει όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία η, η Ευρωπαϊκή Ένωση οπωσδήποτε θα πρέπει ε, να έχει σε αυτόν τον παγκοσμιοποιημένο κόσμο ε, το απαραίτητο, την απαραίτητη δεξαμενή ε, καλά καταρτισμένων ανθρώπων. Αυτή τη στιγμή, ειδικά στην έρευνα, πρέπει οπωσδήποτε να το λάβουμε υπόψη μας. Αυτή τη στιγμή στην έρευνα τουλάχιστον οι γυναίκες είναι πολύ λιγότερες ε, οι προσπάθειες της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας έχουν ως στόχο να υλοποιηθεί σωστά αυτή η προτεραιότητα του οδικού χάρτη. Η Λουξεμβουργιανή Προεδρία θα ήθελε ιδιαίτερος να υπογραμμίσει ε, όλα τα στοιχεία του σχεδίου για την ισότητα των φύλων στα πλαίσια της οποίας θα υπάρχει διαφάνεια, καμία διάκριση ανδρών γυναικών, ε, προσλήψεις που θα βασίζονται στα προηγούμενα, καθώς επίσης και στην πραγματική αριστεία. Με τον τρόπο αυτό θα επιτύχουμε καλύτερη ισορροπία ανδρών και γυναικών στα, στις θέσεις ε, ε, ηγεσία και λήψης απόφασης. Εμείς θεωρούμε ότι σε όλες τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις αυτό το στοιχείο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Ε, στο πέρας της άτυπης συνεδρίασης της επόμενης Τρίτης ενδεχομένως θα μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε τις αρχές αυτές σε κάποια συμπεράσματα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ε, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι η σωστή διακυβέρνηση, καθώς επίσης και ο συμβουλευτικός ρόλος θα αποτελέσουν, ε, ε, θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία της Λουξεμβουριανής Προεδρίας βάσει πάντα των όσων συμφωνήθηκαν την 29η Μαΐου. Ε, ευελπιστούμε ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί υπό δική μας Προεδρία τον Δεκέμβριο τρέχοντος έτους και με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την συμβουλευτική διαδικασία του Ευρωπαϊκού Χώρου μετά από πολλές συζητήσεις και με βάση ε, της ευρείας συνενέσεως ε, που αφορά το θέμα αυτό. Η, η Προεδρία θα δείξει πνεύμα συνεργασίας με, με την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη έτσι ώστε το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας ε, να είναι σε θέση ε, να, ε, να δώσει πράσινο φως για την επαναδιαπραγμάτευση της ΕΡΑΚ, της Συμβουλευτικής Δομής η, επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό ρόλο της ΕΡΑΚ θα της δώσουμε την δυνατότητα να παίξει πλήρως τον ρόλο και ε, την ουσία για την οποία έχει δημιουργηθεί, ε, να δίνει πρώιμες γνωμοδοτήσεις ε, στην Κομισιόν, να αυξήσει την αριστεία και την ανταγωνιστικότητα μέσα από καλύτερο συντονισμό και καλύτερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φορέων και με τον τρόπο αυτό να προωθήσει την έρευνα. Επιτρέψτε μου να περάσω τώρα σε μία άλλη προτεραιότητα της Προεδρίας μας, κύριε Πρόεδρε, δηλαδή την ακεραιότητα της έρευνας. Κανένας από εμά δεν θα αρνηθεί ότι ανάμεσα στην ε, έρευνα, στην ποιοτική έρευνα ε, και την οικονομική ευμάρεια και την πρόοδο ε, ότι υπάρχει διασύνδεση. Ε, και σε τεχνικό, τεχνολογικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο κατανόησης ε, πιστεύουμε ότι πολλά μπορεί να κερδίσουμε από τη βελτίωση της επιστημονικής έρευνας σε όλους τους τομείς ε, αλλά ιδιαίτερως στις STEM τεχνολογικές, οικονομία και μηχανική. Αυτοί είναι οι τομείς οι οποίοι εγγράφονται σε ευρύτερο ε, πολιτικό πλαίσιο βάσει της στρατηγικής 2020. Ε, Πρόκειται για βιώσιμα ε, εργαλεία, συμμετοχικά εργαλεία και νομίζουμε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σωστά απέναντι στους ανταγωνιστές η εγγενής ουσία της γνώσης βασίζεται ε, στο γεγονός ότι οι επιστημονικές γνώσεις είναι ανεξάρτητες, ελεύθερες, ε, χωρίς να έχουν υποστεί οποιαδήποτε οικονομική, πολιτική ή ιδεολογική ε, πίεση. Αυτό μπορεί να φανεί καλύτερα και στα αποτελέσματα της, αποτελέσματα της έρευνας. Αυτό βεβαίως θα έχει στη βάση του την εμπιστοσύνη της κοινή γνώμης στο αποτέλεσμα της έρευνας. Αυτό όμως προϋποθέτει οπωσδήποτε την ακαιρεότητα της έρευνας και εν γέννη της επιστήμης. Γι' αυτό η Λουξεμβουργενή Προεδρία θα προσπαθήσει να οδηγήσει ε, στην, ε, σε αυτήν την ε, αρχική, ε, ε, σε αυτήν την ε, πλήρη εφαρμογή της ακαιρεότητας και της ανεξαρτησίας από την πρώτη σκέψη μέχρι το τελικό προϊόν. Είναι σαφές βεβαίως ότι σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να βοηθηθούμε και από την πρακτική ε, από τις λύσεις των βέλτιτων ε, πρακτικών. Το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ αναφέρει ε, ακριβώς αυτό το θέμα της πρόθεσης της ακαιρεότητας στην έρευνα και την εμπιστοσύνη που αφενός καλούνται να δείξουν ακεραιότητα ενώ αφετέρου να προωθήσουν την διαφάνεια και την δικαιοσύνη σε όλες ε, τις ερευνητικές διαδικασίες. Ε, μία πιο εναρμονισμένη και πιο ε, προενεργητική ε, ε, διατύπωση η οποία θα ξεπεράσει τα εθνικά συστήματα και θα μπορούσε να βοηθήσει ε, γενικότερα την έρευνα. Είναι κοινό αποδεκτό ότι το καλύτερο εργαλείο πρόληψης είναι ενδεχομένως αυτό που μπορεί να οδηγήσει σε καλά αποτελέσματα. Ταυτόχρονα όμως χρειαζόμαστε και ειδική ε, εκπαίδευση προσαρμοσμένη στους ε, ερευνητές ε, και που θα δημιουργήσει την νέα γενιά των ερευνητών. Θέλουμε κατάρτιση η οποία θα είναι σωστή και η οποία καλά θα επηρεάσει, θετικά θα επηρεάσει του, την συμπεριφορά των νέων ερευνητών και επιστημόνων έτσι ώστε να παραγωνιστούν οι εσφαλμένες ε, συμπεριφορές. Ε, θα πρέπει να συζητήσουμε ε, και το θέμα της πρόληψης των ελλείψεων των επιστημονικών έτσι, και αυτό να είναι βασικό στοιχείο των επιστημονικών, της επιστημονικής καριέρας και της ερευνητικής καριέρας. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να παίξουμε καταλητικό ρόλο ε, ασχολούμενοι με την έρευνα έτσι ώστε η πρόληψη αυτής ε, της, ε, αυτών των ελληματικών συμπεριφορών να είναι πλήρης. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολήθηκε με το θέμα της ακεραιότητας της έρευνας στον ορίζοντα 2020 γίνεται σαφής αναφορά στην ακεραιότητα της έρευνας. Η αρχή αυτής της ακεραιότητας στα πλαίσια του ορίζοντα 2020 νομίζω ότι σαφώς αντικατοπτρίζει την άποψη του επιστημονικού κόσμου. Αυτή η συζήτηση της ακαιρεότητας ε, της ε, έρευνας οπωσδήποτε θα φυγεί την επόμενη εβδομάδα στην άτυπη συνεδρίαση του Λουξεμβούργου. Η δε Λουξεμβουργιανή Προεδρία ε, θα ήθελε να εγκριθούν συμπεράσματα από το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας που προβλέπεται να συνεδριάσει την 1η Δεκεμβρίου του 2015. Με τον τρόπο αυτό θα έχουμε πιο ομοιογενοποιημένες και πιο τυποποιημένες αρχές οι οποίες ε, ε, θα αναφέρονται σε, ε, σε όλα τα επιστημονικά προγράμματα. Μπορούμε επίσης να προτείνουμε πιο εναρμονισμένες κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την έρευνα βασιζόμενη στους ήδη υπάρχοντες κώδικες ε, συμπεριφοράς. Ολοκληρώνοντας πρέπει να πω κύριε Πρόεδρε ότι η δράση της Ουκρανικής Προεδρίας εγγράφεται πλε, πλήρως στο πρόγραμμα του Προέδρου της Επιτροπής Jean-Claude Juncker που μπορεί να δημιουργήσει μέσω μοχλεύσεως πάνω από 200 δις ευρώ. Ε, θεωρούμε ότι ε, θα ε, κινητοποιηθούν μέσω του προγράμματος αυτού πολλές δυνάμεις και κονδύλια τα οποία θα αυξήσουν την χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος και θα δημιουργήσουν μεγαλύτερη κινητικότητα. Γι' αυτό λοιπόν προτιθέμεθα στο Συμβούλιο Διαγωνιστικότητα της 1ης Δεκεμβρίου να γίνει ιδιαίτερη συζήτηση για, το, ε, για αυτό το πρόγραμμα στρατηγικής ε, ε, χρηματοδότησης έτσι ώστε από ε, τα 2,2 δις ευρώ του ορίζοντα 2020 και που χρησιμοποιούνται ε, σαν εγγύηση για το ε, επενδυτικό πρόγραμμα της Ευρώπης να τα χρησιμοποιήσουμε λέω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτά ήθελα να σας πω και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Uh, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ για την παρουσίασή σας, εξαιρετικά σαφής και συγκεκριμένη με όλο το χρονοδιάγραμμα των συναντήσεων που έχουμε ενώπιόν μας, που είναι σημαντικό, γιατί πρέπει να προωθούμε συνέχεια την έρευνα και καινοτομία. Τώρα, θα ακούσουμε τις πολιτικές ομάδες. Εξ του ΕΛΚ, ο κύριος Έλερ. Ευχαριστούμε. καλώ ήρθατε στην Επιτροπή μας. Ακούμε τα όσα είπε η Προεδρία για την έρευνα και καινοτομία. Τα ερωτήματά μου είναι πρακτικής φύσεως. Αυτές τις ημέρες, σήμερα και αύριο, καθορίζεται και η ε, γραμμή του Κοινοβουλίου ε, για το 2016 σε ό,τι την καινοτομία. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή backlogging για τον ορίζοντα 2020, όμως μας είπαν ότι το 2016 δεν υπάρχουν ε, όρια για αυτό το είδους το backloading. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή αξιοποιούν 150 εκατομμύρια αυτών των μη υφιστάμενων ορίων για να ε, θεσπίσουν ε, προγράμματα έκτακτη ανάγκη για του πρόσφυγε. Και πολύ σωστά κάνουν. Αλλά πρακτικά πώ το Συμβούλιο και η Επιτροπή λένε ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι στο γενικό αποθεματικό και πώς γίνεται αν ήδη από το 2016 ζητήσουμε ε, αλλά και στη συνέχεια να έχουμε ένα συγκεκριμένο ε, συντελεστή και ποσοστό για τον του 2020. Αυτό είναι το ένα. Μετά. Πώς βλέπετε αυτή τη διαφορά. Αφενός τα διαστατικά ταμεία καλούμε τα κράτη-μέλη όταν θα πανούν τα κονδύλια, το εθνικό ταμείο να τα αξιοποιούν κατά ένα τρίτο για την έρευνα και κοινοτομία να ορίσουν τον στόχο επίτευξη του 3% σε ό,τι αφορά τι ε, γενικέ δαπάνε έρευνα και κοινοτομία και ταυτόχρονα η ίδια Προεδρία, η ίδια Κομισιόν μειώνει την ε, χρηματοδότηση για το R&D κάτω του 2%. Από τη μία λοιπόν ζητούμε να αυξηθεί η χρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη μέσω των Εθνικών Ταμείων και ταυτόχρονα περικόπτουμε τις ε, δαπάνες για την έρευνα και κοινοτομία κάτω από το 2% του ΑΕΠ στην Ευρώπη. Δεν μπορώ να το κατανοήσω αυτό. Ευχαριστώ. Για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, η κυρία Κρέελ. Μάλιστα, σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Μου άρεσε πάρα πολύ το ότι μία από τις πιο σημαντικές προτεραιότητές σας στον ευρωπαϊκό ερευνητικό χώρο είναι η διάσταση των φύλων γυναικών και ανδρών γνωρίζω ότι αυτό το θέμα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωκοινοβούλιο δεν είναι καθόλου εύκολο να συζητηθεί και να προαχθεί. Αλλά γνωρίζω ότι και το ίδιο ισχύει και για το Συμβούλιο. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Η ομάδα μας θα σας παρακολουθήσει και θα σας συνοδεύσει σε αυτή την κατεύθυνση και πορεία. Ζητούμε να υπάρξουν περισσότερες δυνατότητες στην έρευνα. Είναι ένα θέμα λοιπόν όχι μόνο προκηρύξεων και διαφάνειας, σε αυτή την κατάσταση που έχουμε σήμερα, αλλά είναι επίσης ένα θέμα δημιουργίας ευκαιριών, ώστε να είναι συμβατή και να συνάδει η οικογενειακή ζωή με την επαγγελματική ζωή. Αυτό αφορά γυναίκες και άνδρες εξίσου. Γι' αυτό είμαστε πρόθυμοι να σας βοηθήσουμε και να σας ακολουθήσουμε σε αυτή την πορεία. Θα ήθελα ένα σημείο να αναφέρω που αφορά τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Τους τελευταίους μήνες επανειλημμένα Διαρκώς ε, τίθεται το ερώτημα από τους εταίρους μας σε συζητήσεις τι εννοούμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τον Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Χώρο. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που πρέπει να αποσαφινιστούν ως προς τους πολίτες και θα ευχόμουν η Λουξεμβουριανή Προεδρία να συνεισφέρει να υπάρξει σαφήνεια για την έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα προγράμματα και σχέδια να καθοριστούν που μελλοντικά θα, θα τύχουν συνέχειας για το ένα ή άλλο θέμα όπου υπάρχουν κάποιες ασάφειες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω επίσης κάποιες δραστηριότητες προβλέπονται στο πλαίσιο Γαλιλαίου και Κοπέρνικου, Γαλιλαίο και Κοπέρνικους κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Ένα τρίτο θέμα. Είμαι μέλος και στην Επιτροπή Ήτρε αλλά και μέλος της Επιτροπής της Περιφερικής Ανάπτυξης. Και τίθεται το ερώτημα αυτό εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα είχαμε συμφωνήσει όχι μόνο κάποια κονδύλια στον τομέα της έρευνας να διατίθενται, αλλά δημιουργήσαμε και τη δυνατότητα κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο να συνδέονται με τον ορίζοντα 2020, Horizon 2020 Program. Τώρα τα λειτουργικά προγράμματα σχεδόν όλα έχουν εγκριθεί και θα ήθελα η Προεδρία πραγματικά αυτή τη διασύνδεση ορίζοντα 2020 Horizon 2020 και την πολιτική συνοχής να τα παρακολουθήσει ενεργά και εκ του σύνεγγυς και από τα κράτη-μέλη να γίνει αυτή η προσπάθεια και να υπάρξει μεγάλη διάχυση των δραστηριοτήτων για να δούμε πώς τέτοια προγράμματα μπορούν να διαμορφωθούν από κοινού. Διότι θα έλεγα αυτή η διασύνδεση αφενός δημιουργίας υποδομών για την έρευνα συνεργασίας με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και προγράμματα και σχέδια για τον ορίζοντα 2020 είναι πολύ σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούν να μας δώσουν την όθηση για την πρόοδο. Ευχαριστώ για τους συντηρητικούς μεταρρυθμιστές ο κύριος Χένκελ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής μας. Κύριε Υπουργέ, ήμουν επί πολλά χρόνια υπεύθυνο για μια ερευνητική κοινότητα στην Γερμανία που 86 ερευνητικά ιδρύματα έχει στη Γερμανία και 15.000 ερευνητές συνολικά. Και πρέπει να σας πω το χειρότερο που είχα ζήσει είναι η απίστευτη αβεβαιότητα και ανασφάλεια που από τις εθνικές κυβερνήσεις αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχονται. Και θα ήθελα εδώ κάποια πράγματα να αναφέρω. Εν μέρει αναφέρθηκε από πλευρά του κυρίου Ερέφιο Πέιν Πρώτον, οι προσπάθειε ορίζοντα του 2020 να λαιλατηθεί, να απογυμνοθεί. είναι απίστευτε, Δημιούργησαν πολύ μεγάλη δυσφορία, μεγάλη δυσαρέσκεια, διακομματικά. Είναι εντυπωσιακό να δει κανεί ότι τα κόμματα εδώ συμφώνησαν όλα, ότι αυτό ήταν απαράδεκτο. Και κατά τα άλλα έχουμε και πολλές κοινοβουλευτικές επιτροπές που εξοργίστηκαν με αυτή την κατάσταση. Μια τέτοια κατάσταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν την έχω ζήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να συμφωνούν όλοι ότι κάτι είναι απαράδεκτο και δεν έπρεπε να συμβεί. Δεύτερον, <clears throat> η κατάργηση του Chief Scientific Advisor, του κύριου ε, επιστημονικού συμβούλου μας, ανησύχη, μας ανησύχησε και το πώς αντιμετωπίστηκαν αυτά τα θέματα σε σχέση με την Επιτροπή. Τώρα, τι μας προτείνουν. Μια νέα διαδικασία μας υποσχέθηκαν που θα μεριμνήσει λέει και θα φροντίσει να δίνονται συμβουλές και κατευθύνσεις από την scientific community, την επιστημονική κοινότητα. Παρακαλώ θερμά, για κοιτάξτε αυτή τη διαδικασία. Πώς έχει. Είναι πραγματικά ανεξάρτητη η διαδικασία μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα ή μήπως κάποια άτομα ζητείτε να συμμετάσχουν που έχουν κάποιους άλλους σκοπούς που θέλουν να εξυπηρετήσουν. Αυτό ήταν το ενδιαφέρον σε σχέση με την CSA, ότι είχαμε μια επιστήμονα απέναντί μας που το μόνο που την ενδιέφερε ήταν τα επιστημονικά αποτελέσματα και οι επιστημονικοί στόχοι. Το τρίτο ήδη αναφέρθηκε. Μπορώ να πω για τον στόχο του 3% καλό θα ήταν η δική μας αυτή η Προεδρία του Λουξεμβούργου να λέει ότι οι Αμερικανοί ή οι Άπωνες δίνουν πολλά περισσότερα κονδύλια. Επενέστε την Φινλανδία και τη Σουηδία και να ψέξετε όλες τις χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αυτό το στόχο του 3% δεν τον πετυχαίνουν. Και ένα τελευταίο σημείο, το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλές, αλλά θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Έχω την εντύπωση ότι για το αποτέλεσμα μιας ετοιμιγορίας, ενός δημοψηφίσματος, τιμωρούνται κάποιοι σε κάποιο σημείο για το, που δεν είχε κανένα, καμιά σχέση με δημοψήφισμα. Αν τώρα εδώ υπάρχουν υπάρχουν κυρώσεις και αν εμείς στην συνεργασία με την Ελβετία λόγω αυτού του δημοψηφίσματος εμείς την παγώσουμε ή την παρακολύσουμε τη συνεργασία με την Ελβετία, τότε θα αυτοϊπονομευθούμε. Θα είναι εις βάρος μας αυτό. Να υπενθυμίσω ότι το το μεγαλύτερο ερευνητικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα διεξάγεται στην Ελβετία με τον επιταχυντή. Παρακαλώ λοιπόν αυτό εξ ονόματός μας να το λάβετε υπόψη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φεντερικ Φέντερλε από την Άλντε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τον Υπουργό που μας παρουσίασε τις προτεραιότητες. Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο να ακούμε ότι η Προεδρία σας ε, θέλει να ε, θέσει ως προτεραιότητα την έρευνα. Ακούσατε και τους συναδέλφους ότι αποτέλεσε αλλαγή στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά την έρευνα. Και έτσι είναι ενθαρρυντικό ότι και εσείς προτίθεστε να ενισχύσετε την έρευνα σε μια περίοδο που πολύ φοβόμαστε, ειδικά σε αυτή την Ευρώπη, στο, σε αυτή την Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι αποσύρονται και περικόπτονται πόροι και κονδύλια για την έρευνα που είναι απαραίτητη και την καινοτομία για το μέλλον. Είπε ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία λοιπόν στον τομέα της έρευνα και καινοτομία υπό την Προεδρία σα, Είναι σημαντικό γιατί υπήρξε πολύ μεγάλη ανησυχία επειδή υπάρχουν προβλήματα με τα μεγάλα ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω τις εξής σκέψεις. Πρώτον, για την ε, ισότητα μεταξύ των φύλων. Και εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να διορθώσουμε τις ανισορροπίες ό,τι αφορά την κατανομή ε, των ε, πόρων για την έρευνα και η καινοτομία. Και συμφωνώ εδώ με τον σοσιαλιστή συνάδελφο ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δεύτερον, ένα πιο συγκεκριμένο ερώτημα. Μία από τις μεγαλύτερες απειλές προς την ανθρωπότητα είναι το θέμα της αντιμικροβιακής ε, αντοχής που αυξάνεται σε πολλούς ε, τομείς. Ε, βλέπουμε ότι από μια μελέτη που έγινε πριν από 4 χρόνια ήδη 25.000 ζωές χάνονται πρόωρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί πλέον δεν λειτουργούν, δεν πιάνουν αν θέλετε τα αντιβιωτικά. Είναι μια πραγματικότητα και πολύ σύντομα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κατανοήσει ότι ε, οι πολίτες της δεν πρέπει ποτέ να φτάσουν στη σύνταξη, για παράδειγμα. Ε, γιατί πρέπει να κάνουμε κάτι με τα αντιβιωτικά και οι εργοδότες θα πρέπει να αρχίσουν να αγχώνονται γιατί θα πρέπει να βρουν αντικαταστάτες ε, εφόσον οι υπάλληλοι τους θα ε, ασθενούν πιο γρήγορα και θα υπάρχει, είναι τεράστιο οικονομικό κόστος στο μέλλον. Πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο να λύσουμε αυτό το ζήτημα με τα αντιβιωτικά μέσω τη έρευνα, να βρούμε νέα αντιβιωτικά, να έχουμε ένα καθολικό σύστημα και πρόγραμμα για, το, για τις ουσίες που επιτρέπονται για ένα αντιβιωτικό, γιατί ξέρουμε ότι αν βρούμε τώρα ένα νέο αντιβιωτικό, μέσα σε 8 χρόνια θα έχει επέλθει ήδη η αντιμικροβιακή αντίσταση. Με τη δική σα ηγεσία, λοιπόν, θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν πολλέ ενδιαφέρουσε πρωτοβουλίε σε επιμέρου χώρε, όμω αν καταφέρουμε να συλλέξουμε αυτές και να συγκεντρώσουμε αυτές τις δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούμε πολλά περισσότερα να κάνουμε από κοινού. Ευχαριστώ. Κλώτ Τούρμες, εκ μέρου των Πρασίνων. Ευχαριστώ, Τζέζι. Μεγάλη μας χαρά υποδεχόμαστε κι άλλον έναν εκπρόσωπο της κυβέρνησής μου, λέω, γιατί και εμείς συμμετέχουμε ως πράσινοι. Κατά πρώτο θεωρώ ότι η Λεξομβριανή Προεδρία ε, θα τύχει εξαιρετικά καθερμή υποδοχή ε, στο Κοινοβούλιο, επειδή έθεσε ως προτεραιότητα το θέμα της πρόσβασης ε, στις γυναίκες και της διάσταση του φύλου στην ερευνητική πολιτική. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Ένα γενικό σχόλιο μόνο. Όταν συνομιλώ με νέου ερευνητέ, συχνά διαπιστώνω ότι είναι πολύ έντονη η επισφάλεια που προκύπτει από τις συμβάσει τους. Υπάρχει λοιπόν το ζήτημα τη ισορροπία ανδρών και γυναικών, όμω πέραν τούτου πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσο αυτέ οι κακοπληρωμένε συμβάσει ε, που λήγουν μετά από 2-3-5 χρόνια. Υπάρχει και μια γενικότερη, αν θέλετε, διάσταση. Η σταθερότητα δηλαδή που χρειάζεται ένα νέο ερευνητή αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και δεν είναι τυχαίο που στη ΣΥΠΑ και αλλού τα πράγματα είναι καλύτερα. Ίσως πρέπει λοιπόν να διευρύνουμε. Και από αυτή την έννοια χαίρομαι που η Λουξεμβουργιανή κυβέρνηση ήταν μία από, ε, από εκείνες που θέλησαν ε, να επεκταθεί ε, το Marie Curie, ε, αυτή η υποτροφία για τους νέους ερευνητέ. Όμως πρέπει να το εξετάσουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Μετά, σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει για την θεμελιώδη έρευνα, αλλά κατά μία χρονική στιγμή που τίθενται πολλά ζητήματα στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα τη μεταποιητική βιομηχανία, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πρέπει, θεωρώ, να δούμε πώ μπορούμε να οικοδομήσουμε και να διαμορφώσουμε μια καλύτερη ανταλλαγή πέραν των συνόρων για την εφαρμοσμένη έρευνα. Έχουμε εξειδικευμένα Ινστιτούτα για την καινοτομία. Πώς λοιπόν σε αυτούς τομείς μπορούμε να προχωρήσουμε. Βεβαίως δεν θα είναι εύκολο αυτό, γιατί κάθε κράτος μέλος ταυτόχρονα όταν υπάρχει έρευνα που είναι κοντά στην αγορά, περιμένει να έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα και να διατηρήσει για την ίδια ε, τα ωφέλη. Μπορούμε όμως να επιτρέψουμε κάτι τέτοιο απέναντι στους γίγαντες όπως είναι η ΕΠΑ και η Κίνα. Μπορούμε να επιτρέψουμε αυτά τα εθνικά στεγανά σε ό,τι αφορά ε, την έρευνα και την καινοτομία. Σε ό,τι αφορά την ακαιρεότητα, εντάξει δεν χρειάζεται να επεκταθώ. Νομίζω ότι χωρίς ακαιρεότητα θα χαθεί και αξιοπιστία της έρευνας. σα θα το αναφέρατε. Και τέλος, και ο συνάδελφος Χένκελ και ο κύριος Άιλα. όλοι βλέπουμε αυτή την ε, πρόταση αρνητικά το να πάρουμε δηλαδή χρήματα από την έρευνα. Πρέπει τουλάχιστον να διασφαλίσουμε ούτως ώστε το επενδυτικό πρόγραμμα Juncker να δίνει πραγματικό κίνητρο για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλες να χρηματοδοτήσουν ε, τις ερευνητικές υποδομές. Και νομίζω ότι τα όσα είπε η κυρία Κρέλ και η γέφυρα μεταξύ του ορίζοντα 2020 και των διευθυντικών ταμείων θα πρέπει να ενισχυθεί ε, η διασύνδεσή τους με το πρόγραμμα Juncker. Γιατί έχουμε να συνδυάσουμε τα διευθυντικά ταμεία, τα καινοτόμα χρηματοπιστωτικά μέσα για να επενδύσουμε στις υποδομές. Εκεί είναι το κλειδί της μεγαλύτερης απόδοσης. Και νομίζω ότι κατά τη διάρκεια της ε, προεδρίας μας και σε αυτή τη διάσκεψη την 1η Δεκεμβρίου θα πρέπει πραγματικά να συζητήσουμε αυτό το σημείο, να εξετάσουμε σε βάθος τα προγράμματα που βασίζονται στα διαστατικά ταμεία και να δούμε κατά πόσο το ΕΦΣΙ, το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, μπορεί να βοηθήσει περαιτέρω. Και καλά κάνουμε και τις ανασχετούμε με το να αφαιρεθούν πόροι από την έρευνα. Πρέπει να προσέξουμε πολύ, ούτως ότι τουλάχιστον τμήμα αυτών των χρημάτων να επανέλθει στην έρευνα και κοινοδομία. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Είναι πολύ καλέ μέρε για σένα, Κλοντ. Πολύ καλή μέρα σημερινή, γιατί μιλάς περισσότερο από τον οποιονδήποτε άλλο, όπως βλέπεις. Γιατί είσαι στην καρδιά της Ευρώπης, όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά και πνευματικά, γιατί εκπροσωπείς την Προεδρία. Μέχρι το Δεκέμβρη βέβαια θα πάει αυτό. Ναι, το Δεκέμβριο ξαφνικά θα σταματήσω τα πάντα. Θα με επαναφέρετε στον ε, κανονικό χρόνο ομιλίας. Σας ευχαριστώ που μας υπενθυμίσετε και το πρόγραμμα Curie, πολύ σημαντικό για όλους μας. Η κυρία Κάπελ, εξ του ΙΕΝΕΦ. E Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υφυπουργέ, με εντυπωσιάσατε πολύ σήμερα που είπατε ότι στο Λουξεμβούργο οι δημόσιες δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη κατά τα τελευταία 15 χρόνια από 27 αυξήθηκαν σε πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ. Δωδεκαπλασιασμός των δαπανών. Και αυτό σημαίνει ότι ετήσια 1% κατά αυξήσατε τα κονδύλια. Δεν πρέπει άλλες χώρες εδώ να επενέσουμε. το Λουξεμβούργο έχει το best practice, την βέλτιστη πρακτική εδώ και είναι πρωταθλητής όσον αφορά την έρευνα και ανάπτυξη πανευρωπαϊκά. Κύριε Υφυπουργέ, μας, είπατε ποια είναι τα κέντρα βάρους ε, από πλευρά της Λουξεμβουριανής Προεδρίας. Η συνέχιση για την κατεύθυνση του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας ολοκληρωμένη έρευνα. Ευχαριστώ που είπατε ότι τον διοντολογικό κώδικα θέλετε πολύ γοργά να τον εγκρίνετε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την ε, δραστηριότητα στην έρευνα. Και το τρίτο, η βέλτιστη διασφάλιση των θεμάτων των φύλων και η θεσμική διαφύλαξη της ισότητας. Είναι καλό λοιπόν και το διάβασα και αν δει κανείς τις μελέτες αυτές τότε θα διαπιστώσει ότι οι γυναίκες σε ηγετικέ θέσεις είναι αυτό που λείπει και αν υπάρχουν, αν υπήρχαν τέτοιες δυνατότητες να έχουν ηγετικέ ε, θέσεις οι γυναίκες θα είχαν καλύτερες ευκαιρίες και θα είχαν και μια δυνατότητα να βρεθούν στην πρώτη κατηγορία όσον αφορά αυτό σε εισαγωγικά το πρωτάθλημα και η Λουξεμβουργική έγινε η αρχή με την advisory, δηλαδή συμβουλευτική διαργασία και μας είπατε μέχρι το Δεκέμβριο θα υπάρξει μια πρόταση από πλευρά σας για το τι θα γίνει σε σχέση με τις κατευθύνσεις. Αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για την έρευνα και τις επιστήμες, είναι σημαντικό και η επιχειρησιακή πείρα και η υλοποίηση των τεχνολογικών και επιστημονικών πορισμάτων και συμπερασμάτων να λαμβάνονται υπόψη. Ερώτησή μου, ποια βήματα ή διαβήματα θα κάνετε ή έχετε αρκετά στελέχη από τον επιχειρησιακό τομέα και την εφαρμοσμένη έρευνα αυτή την διακυβέρνηση να την διασφαλίσετε ώστε και οι επιχειρήσεις και η πρακτική μορφή να συνδυάζεται και το άλλο το οποίο αναφέρθηκε στο πρώτο, στην πρώτη συνάντηση που είχαμε σήμερα το πρωί με τον Πρωθυπουργό Μπέτερ, η ψηφιοποίηση, κέντρο βάρους της Λουξεμβουριανής Προεδρίας και αυτό είδα να απουσιάζει το κέντρο βάρου στην έρευνα και ανάπτυξη σε σχέση με την ψηφιοποίηση. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα για την ψηφιοποίηση. Είναι ένα εξαιρετικό θέμα, ευρύτατο, όσον αφορά την έρευνα και την αποκεντροποίηση μέσα στο ίδιο το πλαίσιο της ψηφιοποίησης. Για μια διάσκεψη που θα γίνει, θα ε, εξεταστούν αυτά τα θέματα. Η δεύτερη μου ερώτηση προς εμάς είναι Πώς θα διασφαλίσετε κονδύλια για την έρευνα και ανάπτυξη όσον αφορά την ψηφιοποίηση. Ποια συγκεκριμένα μέτρα και πρωτοβουλίες προβλέπετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά από τις πολιτικές ομάδες και τώρα μπορούμε να δώσουμε το λόγο σε μεμονωμένα μέλη. κυρία Ντυρκούνεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ ως μεμονωμένη ευρωβουλευτής μπορώ να πάρω το λόγο. Σας ευχαριστώ τον κύριο Χάντσαν για την παρουσίασή του. Το Λουξεμβούργο μπορεί να είναι μικρή χώρα σε ό,τι φορά την έρευνα για καινοτομία, όμω ε, αποτελεί καλό παράδειγμα για όλου μα, γιατί ξέρω ότι είστε ιδιαίτεροι δραστήριοι και οι φοιτητέ σα στο Λουξεμβούργο. Περίπου 30% συμμετέχουν ε, σε κάποιο, κάποιες κατηγορίες ε, πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών όπως τα Erasmus και το καθεξής και αυτό είναι πολύ σημαντικό παράδειγμα για όλους. Πρέπει να ενθαρρύνουμε όλους τους φοιτητές ανά την Ευρώπη να συμμετέχουν στα προγράμματα όπως το Erasmus. Επικεντρώνωστε σε καλά στοιχεία, θεωρώ, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Η είσοδο των φίλων είναι εξαιρετικά σημαντικό θέμα και καλό είναι που θέλετε να ενθαρρύνετε τις ε, ταλαντούχε γυναίκες να να συνεχίσουν ε, τη σταδιοδρομία τους. Πράγματι πολλά έχουμε ακόμα να κάνουμε σε αυτό το τομέα και θετικό είναι επίσης ότι επικεντρώνεστε στην ε, βασική θεμελιώδη έρευνα γιατί πρέπει να ενισχυθεί αυτή η έννοια της θεμελιώδη και της ευρωπαϊκής έρευνα. Γιατί αν δείτε τα κύρια, τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, δεν είναι πολλά από την Ευρώπη. Τα 20 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου είναι περίπου 4 ενδεχομένως της Ευρώπης, τα υπόλοιπα είναι τον ΙΠΑ. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση. Ήδη αναφέρθηκε προηγουμένως σε όλους τους προβληματισμούς που έχουμε με το πρόγραμμα Horizon 2020. Είναι κάτι που μας απασχολεί ιδιαίτερως και πάντα μας ε, προβληματίζουν οι περικοπές ε, στον προπολογισμό αυτού του σημαντικού προγράμματος. Είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στη βασική έρευνα, αλλά από την άλλη έχουμε και το θέμα της, την πλευρά της, ε, της επιχειρηματικότητας, γιατί έχουμε καλές ιδέες στην Ευρώπη παραδοσιακά, αλλά δεν τα πάμε καλά όταν πρέπει να το μεταφέρουμε αυτό στην πράξη. Δεν ξέρω τι σχεδιάζετε να κάνετε σε ό,τι αφορά την καινοτομία και σε σχέση με τις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ κύριο Στοσανόφσκι. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό. Πολύ θετικό είναι που η Προεδρία του Λουξεμβούργου ασχολείται με το σημαντικό θέμα της έρευνας και Κατανοείται ότι η ποιοτική έρευνα και η ε, μετάφραση της καινοτομίας, της έρευνας μάλλον σε καινοτομία, είναι από τα βασικά στοιχεία της ανταγωνιστικότητας των κρατών μελών. Και χρειαζόμαστε την έρευνα σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας και της Ενεργειακής Ένωσης. Γιατί χωρίς αυτή την έρευνα δεν θα έχουμε τις ε, απαραίτητες λύσεις. Εγώ για πολλά χρόνια είμαι ενεργός στο πανεπιστήμιό μου και όπως έχει ήδη υπογραμμιστεί, θεωρώ και εγώ ότι η ισότητα μεταξύ των φίλων είναι κάτι σαν παρενέργεια. Πρέπει και εμείς λοιπόν να μεριμνήσουμε ότως ώστε οι νέοι ταλαντούχοι ερευνητέ να έχουν επαρκή δικαιώματα σε ό,τι αφορά την κοινωνική ασφάλιση αλλά και σταθερότητα στο εργασιακό τους περιβάλλον. Είναι κρίσιμη σημασία για την Ευρώπη το πώς αντιμετωπίζουμε τέτοια ταλέντα. Είτε είναι άντρε είτε γυναίκε, εγώ δεν κάνω διάκριση. πώ θα τα κρατήσουμε αυτά τα ταλέντα, πώ ε, θα διαμορφώσουμε ένα επαρκές, ευνοϊ, επαρκώς ευνοϊκό περιβάλλον, γιατί οι νέοι έχουν και άλλες υποχρεώσεις οικογενειακές ή άλλες. Και θα ήθελα να συμφωνήσω με τους αδέλφους που είπαν ότι όλοι έχουμε παλέψει για τη χρηματοδότηση του προγράμματος Horizon 2020 και μου προκαλεί έκπληξη ότι τώρα ξαφνικά περικόπτεται αυτός ο προπολογισμό. Και έχουμε άλλες προτεραιότητες. Και λέμε ότι δεν ξέρουμε ούτε καν πότε θα επιστρέψουν αυτά τα χρήματα. Κάτι το οποίο δεν άκουσα στην αρχική σας εισήγηση, το οποίο αφορά ε, τα ταλέντα και τον ορίζοντα 2020. Συνεχώς συγκρινόμαστε με την Αμερικανική έρευνα. Σε ό,τι αφορά το equity financing είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ευχαριστώ κύριο Γκύρικ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε στις διαφορετικές προτεραιότητες της Προεδρίας σας για το επόμενο εξάμεινο. Πρέπει να πω ότι μου αρέσουν διότι αφορούν κεντρικά ζητήματα. Όμως και κάτι άλλο, ένα άλλο θεμελιώδες θέμα θα πρέπει να τύχει προτεραιότητας. Ίσως είναι κάτι που θα έπρεπε να ήταν ήδη προτεραιότητα, ήδη κάποιο χρόνο προηγούμενα. Κάνω λόγο εδώ για μια ομάδα ερευνητών σε σχέση με θέματα ασφάλειας. Γνωρίζουμε ότι στον ορίζοντα 2020 αυτό το στοιχείο είναι κάτι το οποίο καλύφθηκε, υπήρξε μια ομάδα επιστημόνων που θα παρακολουθούσαν τέτοιου είδους θέματα και υπήρχαν και όμως και κάποια θέματα τα οποία δεν είχαν επιληθεί. Θα έλεγα ότι ίσως αυτό θα έπρεπε να είχε συμπεριληφθεί ως ε, θέμα και μάλιστα από την τρέχουσα Προεδρία. Διότι βλέπουμε ότι ο σημερινός κόσμος δεν είναι ένας ιδιαίτερα ασφαλής κόσμος. Χρειάζεται λοιπόν έρευνα για την ασφάλεια. Είναι κάτι αναγκαίο σε, μια ε, σε ένα τέτοιο πεδίο για την άμυνα. Ίσως θα έπρεπε να ιδρυθεί, να δημιουργηθεί ένα ίδρυμα για την άμυνα και την ασφάλεια μέσα στο πλαίσιο ακριβώς του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Κέντρου και κάπως να ενταχθεί για να μπορέσει να λειτουργήσει. Αυτό πρέπει να καλυφθεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ματέ παρακαλώ, επόμενος αγορητής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, δεν είμαι από το Λουξεμβούργο, αλλά είμαι από το Ντιονβίλη. Είμαστε γείτονες, κοντά σας. Ε, από σήμερα το πρωί άκουσα τον κύριο Μπέτελ, ε, άκουσα και τον Υπουργό ε, Απασχόλησης ε, που, του Λουξεμβούργου που είχαν πραγματικά μια πάρα πολύ δυναμική, ένα πολύ δυναμικό λόγο πώς μπορούμε να ξαναστήσουμε στα πόδια στην Ευρώπη, την Ευρώπη της τεχνολογίας κτλ. Ε, λυπούμε, ίσως εγώ τώρα θα χαλάσω λίγο τη διάθεση όλων και το ε, την ατμόσφαιρα, αλλά έχετε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία που μας οδηγούν να πούμε ότι αυτή η ε, Ευρώπη της έρευνας και της καινοτομίας ε, έχει βρει το σωστό της βηματισμό και θα προχωρήσει, γιατί δυστυχώς αυτό που βλέπουμε είναι έρχονται και φεύγουν οι προεδρίες, ακούγονται διάφορες ιδέες, αλλά σε κάθε τέλος εξάμηνης προεδρίας ε, μας μένει μία πικρή αίσθηση ότι δεν έχουν γίνει αυτά που είχαν προαναγγελθεί. Ε, θέλουμε να ξεκινήσει η Ευρώπη. Έχετε κάποια στοιχεία να μας δώσετε. Σας ευχαριστώ συνάδελφε. Θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο. Όχι. Επομένως κύριε Υπουργέ, δώστε μας τις ε, απαντήσεις σας. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε την δυνατότητα να απαντήσω στα σχόλια και τις παρατηρήσεις και ερωτήσεις που ακούσαμε. Και βεβαίως εδώ θα ήθελα να χαιρετήσω και τους ε, γείτονες ε, αλλά και τον Κλοντ, αγαπητέ Κλοντ και τον, ε, τους συμπολίτες μου. Ευχαριστώ βεβαίω και όσου ε, πήραν το λόγο έτσι ώστε να κάνουν κάποιο σχόλιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η Προεδρία να έχει γνώση των απόψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, ε, σα βεβαιώ ότι τα στοιχεία τα οποία μας δίνετε και μας υποβάλλετε λαμβάνονται υπόψη και θα ληφθούν στη διάρκεια τη Προεδρία. Υπάρχουν διάφοροι όροι για να να μιλήσουν και, ε, ε, ε, για αυτό που συμβαίνει. Άλλοι λένε λαιλάτιση, άλλοι λένε ε, βάζουμε χέρι στο κορβανά της έρευνας και της τεχνολογίας και θα ήθελα να βγάλω το καπέλο της ουδετερότητας ε, της Προεδρίας και να σας πω ότι εμείς ως Λουξεμβούργο πραγματικά ε, ανησυχούμε, δεν θέλουμε ε, κανένας να βάλει χέρι σε αυτά τα χρήματα και σας υπογραμμίζω ότι εμείς γι' αυτό ακριβώς έχουμε προβλέψει την ανταλλαγή απόψεων τον Δεκέμβριο και υπάρχει και μια ομάδα εργασίας σε επίπεδο ΕΡΑΚ που ε, έχει σαν κύριο στόχο ακριβώς να δει ε, τα όσα έχουν γίνει στις διάφορες επενδύσεις. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί έτσι ώστε τα χρήματα αυτά πραγματικά να επενδυθούν στην έρευνα και την καινοτομία. Ε, προτείνω λοιπόν να περιμένουμε λίγο αυτήν την ανταλλαγή απόψεων η οποία έχει προβλεφθεί να γίνει την 1η Δεκεμβρίου και μετά να κρίνουμε. Επίσης, Καταλαβαίνω την κυρία Κέλ, τον κύριο Φέντερ, την κυρία Καπέλ, την κυρία Βερκούνεν, τον κύριο Τοσανόφσκι που ε, μας στηρίζουν σε αυτήν την προσέγγιση μας όσον αφορά την ισότητα των φίλων και τους ευχαριστώ γιατί πρόκειται για ένα ε, θέμα πολύ σημαντικό. Το έχουμε βάλει στην ημερήσια διάταξη και πιστεύω ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα πρέπει να συζητηθεί μονάχα στα πλαίσια της Λουξεμβουριανής Προεδρίας αλλά και όλα τα επόμενα χρόνια. Κύριε Χέγγελε, να σας απαντήσω. Η Ελβετία ε, θα μπορεί να συμμετάσχει στον πρώτο πυλώνα της αριστείας που είναι ε, ένα από τους προβληματισμούς που εκφράσατε. Και ο κύριος Τούρμες επίσης ε, προβληματίστηκε για την ανταλλαγή ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τον επιχειρηματικό κόσμο και τον ερευνητικό κόσμο. Πρέπει να σας πω ότι στον ορίζοντα 2020 ε, ε, ε, υπάρχει τέτοια σχετική αναφορά. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί και σε εθνικό επίπεδο και λέμε ότι θα πρέπει να προωθηθεί η συνεργασία αυτή αν θέλουμε να έχουμε καλό οικονομικό αντίκτυπο. Επίσης, θα ήθελα ε, να σας ευχαριστήσω κύριε Μαρτάν για τα όσα ε, μας ε, είπατε και είμαι βέβαιος ότι στη διάρκεια της Προεδρίας, της Προεδρίας θα έχουμε την δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις και το προβληματικό του κ. Ένερ επίσης ε, θα την ε, μεταφέρω γιατί βεβαίως ε, δεν είναι δικό μου ζήτημα δικιά μου αρμοδιότητας. Θα την μεταφέρω στον Υπουργό Οικονομικών του Λουξεμβούργου έτσι ώστε να εμφανιστεί και στον προϋπολογισμό το θέμα αυτό. Η κυρία Κρέλ επίσης έθεσε το ερώτημα του προγράμματος Γαλιλαίος δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα. Ε, ο κύριος Σνάιντερ, ο αναπληρωτή Πρωθυπουργό, ε, είναι αυτός ο οποίος παρακολουθεί το θέμα στενά και νομίζω ότι το έχει εγγράψει στην αυριανή ημερήσια διάταξη και επομένως θα μπορέσετε να τον ρωτήσετε ε, για όλα τα στοιχεία τα οποία θέλετε έτσι ώστε να έχετε μια έγκριτη απάντηση. Αυτά ήθελα να σας πω, νομίζω ότι δεν μακρηγόρησα. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τα παρόντα μέλη της Επιτροπής για την ανταλλαγή απόψεων, για το input το οποίο μας δώσατε. Είναι τροφή για σκέψη και ε, βεβαίως νομίζω ότι και ευελπιστώ σύμφωνα και με αυτά που είπε και ο κύριος Μαρτά ότι στο τέλος της ε, Λουξεμβουργικής Προεδρίας η αποτίμηση θα είναι θετική. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ λέει ο Πρόεδρος κύριε Υπουργέ για την ε, παρουσίασή σας. Πρέπει να σας πω ότι τα θέματα τα οποία θίξατε αποτελούν μεγάλη προτεραιότητα της Επιτροπής Ήτρε γιατί θέλουμε τελικά να επιτύχουμε κάτι, ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα το οποίο θα μας βοηθήσει να φύγουμε, να βγούμε από την κρίση. ε, πρέπει να είμαστε πολύ πιο καινοτόμοι, να ξεπεράσουμε αυτό το 2,5-3% του, του ΑΕΠ. Ο τομέας ICT έχει βέβαια και μικρές επιχειρήσεις, μικρομεσαίες, αλλά και η ενέργεια είναι πάρα πολύ σημαντική. Τώρα οδεύουμε προς τη συμφωνία TTIP. Και έχουμε τέτοιες ε, τιμές ε, στην ενέργεια που πραγματικά προβληματιζόμαστε. Επομένως, ε, καινοτομία, ε, ε, πολιτική διαστήματος, όλα αυτά μας απασχολούν πολύ στην Επιτροπή μας. Και χαίρομαι που απασχολούν και εσάς. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα για το επόμενο εξάμεινο. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Uh, dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι. Uh, Mr. Commissioner Ο κύριος uh, Επίτροπος Αρίας Κανιέτε βρίσκεται ήδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά δεν μπορεί να έρθει ακριβώς τώρα. Ε, για τα επόμενα 15 λεπτά τουλάχιστον δεν θα είναι μαζί μας. Ah, ε, να κάνουμε ένα διάλειμμα για καφέ κερασμένο από τον κύριο Αρία Κανιέτε. Κοιτάξτε, θα είμαι ειλικρινή μαζί σας. Έχω εδώ μια σύντομη πληροφόρηση. Ο κύριος επίτροπο Κανιέτε είναι μπλοκαρισμένος στην Επιτροπή Envy. Blocked in Envy Committee λέει το μηχάνημα. Επιτροπή Envy, Επιτροπή Περιβάλλοντος. Τον έχουν μπλοκάρει εκεί. Δεν θέλω να πω τίποτα επιθετικό, δεν θέλω να επιτεθώ στο περιβάλλον, αλλά νομίζω ότι καλό είναι να περιμένουμε 15 λεπτά. Επομένως, διακοπή 15 λεπτά.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 me any Εδώ Ο Επίτροπος κοντεύει να φτάσει στην αίθουσα. Είναι στην τελική ευθεία. Τον περιμένουμε λοιπόν σε ένα-δύο λεπτά. Καθίστε παρακαλώ για να ξεκινήσουμε αμέσως. Dear colleagues, ladies and Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε και κύριοι. Ο Επίτροπο κλιματική ενέργεια και δράση και ενέργεια, μάλλον, ο κύριο Αρια Κανιέτα είναι μαζί μα Μετά από μια δύσκολη συνεδρίαση στην Επιτροπή Περιβάλλοντο από ό,τι ακούω, εμείς πάντως ήπιαμε ένα καφέ στην υγειά σας, κύριε Επίτροπε. Ας περάσουμε τώρα λοιπόν στις σημαντικές συζητήσεις για την διασυνδεσιμότητα και το λιανεμπόριο, ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο. Και όπως ξέρετε σήμερα υιοθετήθηκε το Summer Package με δύο ανακοινώσεις. Μία για την ε, αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, πολύ σημαντικό, αλλά ακόμα πιο σημαντικό ενδεχομένω ανακοίνωση για το New Deal σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές ενέργειας στην Ευρώπη. Ξέρετε κάτι σημαντικό και ενδιαφέρον ζήτημα και θα θέλαμε ε, να σας δώσουμε τώρα το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Ευρωβουλευτέ, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, συγγνώμη για την καθυστέρησή μου. Ήταν περίπλοκες οι εργασίες, έπρεπε να εγκριθεί αυτό το πακέτο στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή και ζητήθηκε να έρθω σήμερα εδώ να παρουσιάσω το πακέτο ενεργειακών μέτρων την πρότασή μα πω θα συμμεθεί πρόοδο για τους κλιματικού στόχους και την αλλαγή των ενεργειακών στόχων. Το καλοκαιρινό πακέτο έχει τι εξή προτάσει. Μια διαβούλευση ε, δεύτερον, μια δυνατότητα να δοθούν αρμοδιότητες στους καταναλωτές, ε, η διαμόρφωση της αγοράς και οι συναφής δράσης. Ξεκινώ με τις ανακοινώσεις ε, σε σχέση με το μέλλον της ενεργειακής αγοράς. Πριν από λίγα χρόνια σε σχέση με τα ανανεώσιμα που ήταν ένα πολύ μικρό περιθωριακό ποσοστό και οι καταναλωτές δεν είχαν ρόλο να διαδραματίσουν στο ενεργειακό σύστημα όσον αφορά αυτά τα ζητήματα. Σύστημα, σήμερα έχουμε ριζοσπαστική αλλαγή των πραγμάτων. Μεγαλύτερη αποκεντρωμένη παραγωγή με όλο και περισσότερες δυνατότητες ευέλικτης ε, ζήτησης καθώς επίσης και την εκπροσώπηση 50% αυτών των δυνατοτήτων παραγωγής μέχρι το 2030 καθώς επίσης και διασυνδεδεμένες αγορές προς όφελος των καταναλωτών. Και πρέπει να αυξήσουμε τις προσπάθειές μας να ανταποκριθούμε σε αυτή τη νέα πραγματικότητα και να μπορέσουμε σε σχέση με τις δυνατότητες να υποφεληθούμε από αυτές. Μια νέα αγορά θα μας δώσει τη θέση να υποφεληθούμε από όλες τις ευκαιρίες που γνωρίζουμε ότι μπορεί να μας προσφέρει αυτή η ενέργεια. Ο ανταγωνισμός είναι η αρχή με την οποία οι επιχειρήσεις μας μπορούν να είναι αποτελεσματικές στον ανταγωνισμό. Η κοινωνική ρύθμιση θα είναι είναι κανόνας και όχι εξαίρεση και οι καταναλωτές θα διαδραματίζουν θετικό ρόλο ως ενημερωμένοι καταναλωτές. Συνολικά μια ολοκληρωμένη αγορά για την ενέργεια που θα δίνει ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης. Αυτή θα είναι η πιο αποτελεσματική δυνατότητα να διασφαλίσουμε τις ενεργειακές μας ε, ανάγκες, ε, την διαμόρφωση της αγοράς και την αντιμετώπιση των κυριότερων προκλήσεων σύντομα να αναφέρω κάποια από τα πιο σημαντικά από αυτά τα στοιχεία. Η συγκεκριμένη σχέση με τα ανανεώσιμα. Έχουμε κάνει μεγάλα άλματα και βήματα και άλματα για την ανταγωνιστικότητα σε αυτόν τον τομέα. Πρόκληση τώρα είναι να εντάξουμε όλα αυτά τα βήματα στην αγορά ενέργειας σας και την, το ηλεκτρικό ρεύμα και σε σχέση με την κατανάλωση αν θέλουμε να επιτύχουμε τους στόχους του 2030 τα ανανεώσιμα θα πρέπει να είναι το ίμιση, το μισό της παραγωγής είναι απόλυτα σαφές λοιπόν ότι αυτό θα αλλάξει σε βάθος το σύστημά μας πολύ περισσότερο από ό,τι είχαμε προβλέψει. Οι διαδικασίες που ξεκινούν θα αλλάξουν τους ε, κανόνες και κανονισμούς για τη μεταβατική αυτή περίοδο. Για να διασφαλίσουμε ότι θα γίνει αυτό πρέπει να βρεθούμε κοντά στους καταναλωτές. Αυτό απαιτεί να κάνουμε τις αγορές πιο ελαστικές, πιο ευέλικτες για να υπάρχει μια ολοκληρωμένη δυνατότητα μέσα σε αυτές τις αγορές να ανταγωνίζονται οι παραγωγοί ε, προς όφελος των καταναλωτών. Θα δίνεται συγκεκριμένη υποστήριξη που θα είναι προς όφελος των καταναλωτών και θα μας δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να στοχεύουμε στις αγορές και να μειώνονται οι στρεβλώσεις των αγορών. Επιπλέον θα πρέπει να γίνει η πραγματικότητα αυτή στην αγορά μια χειροπιαστή πραγματικότητα θα χρειαστούμε λιγότερο δαπανηρές ε, δυνατότητες για να παράξουμε όλη αυτή την ενέργεια. Θα υπάρξουν 100 δις ε, για επενδύσεις χρειαζόμαστε πολύ ε, πιο ε, αποτελεσματική ολοκλήρωση της αγοράς. Η συνεργασία και η συνέργεια πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να πλησιάσουμε ένα ευρωπαϊκό grid, σύστημα διασύνδεσης και δίκτυο. Γι' αυτό πρέπει η ικανότητα των ε, λειτουργών, των παρόχων να αυξηθεί. Οι δυνατότητες λήψης απόφασης και παρεμβάσεων πρέπει να αυξηθεί για την κάλυψη της ζήτησης. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα μέσω μηχανισμών που θεωρούν αναγκαίους τα κράτη-μέλη για την ενεργειακή ασφάλεια. Το μήνυμά μας προς τα κράτη-μέλη σε αυτό είναι σαφές. Συγκεκριμένοι μηχανισμοί δεν είναι αποδεκτοί αν ο στόχος είναι απλά και μόνο να καλύψουν κάποιες απώλειες. Μπορούν να δικαιολογηθούν μόνο αν υπάρχει αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου προβλήματος ε, και δημιουργία δυνατοτήτων. Η αξιολόγηση ενός προγράμματος και η λύση δεν μπορεί να είναι καθαρά εθνικού χαρακτήρα. Πρέπει να είναι ευρωπαϊκού χαρακτήρα ή τουλάχιστον περιφερειακού χαρακτήρα στο τέλος ε, θα πρέπει η ε, εσωτερική αγορά να μετακινηθεί πάλι στο επίκεντρο των πραγμάτων. Ένα σύστημα υποστήριξης θα πρέπει να έχει στόχο τα ανανεώσιμα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα πρέπει να είναι υπό την λειτουργία των, της αγοράς. Και αυτό με οδηγεί στην ανακοίνωση. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι ψηφιακές εξελίξεις προσφέρουν νέες δυνατότητες στους πολίτες ώστε να υποφεληθούμε στα ενεργειακά συστήματα. Εκατομμύρια νοικοκυριά εξαρτώνται από μια παλαιά τεχνολογία θα είναι απλό στην ψηφιακή τεχνολογία να μπορέσουμε με τα ηλεκτρονικά μέσα να σημειώσουμε πρόοδο. Για την κατανάλωση θα υπάρξουν και νέες δυνατότητες δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Η εσωτερική αγορά θα δώσει αυτή τη δυνατότητα με ένα νέο σύμφωνο, New Deal, για τους καταναλωτές. Θα πρέπει ο ρόλος αυτός να ενδυναμωθεί στην Ελλάδα. Θα συνεργαστούμε με ρυθμιστικές εθνικές αρχές, ώστε κάθε πολίτης Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει πρόσβαση σε ένα πιστοποιημένο το σύστημα τιμών ως εργαλείο. Θα μπορέσουμε με δυναμικές συμβάσεις τιμών να ε, ωφελήσουμε τους καταναλωτές και θα εξοικονομήσουμε 30% των δαπανών από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και θα δείξουμε στους πολίτες ότι θα υπάρχει δυνατότητα παραγωγής και κάλυψης των ενεργειακών τους αναγκών. Και έτσι θα πρέπει εκείνοι που δεν χρησιμοποιούν ή δεν θα χρησιμοποιήσουν ε, ε, κάποιο ποσοστό θα επιστρέφεται στο δίκτυο. Και έτσι θα αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα. Το κύριο, μέσο, ε, το κύριο μήνυμα ποιο είναι. Αυτά τα συστήματα ενέργειας να ενταχθούν με αποτελεσματικό κόστος σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ένα εγχείρημα που θα δίνει απαντήσεις σε κάποιες από τις πιο πιεστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Αυτές οι απαντήσεις θα τεθούν μέσα σε συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις, σε προτάσεις κατά το δεύτερο ήμιση του 2015. Ευελπιστώ ότι θα είσαστε δραστήριος παίκτη και θα εμπλακείτε σε αυτό και προσβλέπω στο διάλογο μαζί σας στους επόμενους μήνες. Αγαπητοί συνάδελφοι, ανάφερα τα κυριότερα στοιχεία του πακέτου και θα ήθελα να επικεντρωθώ τώρα στην αναθεώρηση και του ε, συστήματος ε, ε, για την ενεργειακή πιστοποίηση είναι οι προτάσεις που υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προστασία του κλίματος και τις κλιματικές αλλαγές. Θέλω να αρχίσω με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Ρήπων. Η πρόταση που υποβάλλουμε σήμερα είναι μια ανταπόκριση στις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές που υιοθετήθηκαν τον Οκτώβριο 2014. Λιγότερο από 9 μήνες πριν συμφώνησαν οι Ευρωπαίοι ότι πρέπει να μειωθούν οι εκπομπές ρήπων κατά 40% το 2030 και 43% θα γίνει μέσω του συστήματος εμπορίας τρύπων. Αυτό το σύστημα εμπορίας τρύπων κατέδειξε την αξία του κατά το παρελθόν. Σήμερα πρέπει να δείξουμε ότι είναι καλύτερο και πιο αποτελεσματικό. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στις κυριότερες πτυχές αυτής της πρότασης που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Αναφέρομαι στην καλύτερη προστασία όσον αφορά τον άνθρακα και την διαρροή άνθρακα καθώς επίσης και σε στενή συνεργασία σε σχέση με παραγωγές με την παραγωγή. Το ε, σημείο κίνηση είναι ότι κάποιοι τομεί ε, αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο απώλεια ανταγωνιστικότητα στο διεθνέ επίπεδο. Πρέπει να συνεχίσουμε σε σχέση με τι διατάξει διαρροή άνθρακα που θα εκπνεύσουν το 2020 υπό τη σημερινή νομοθεσία, στο σημερινό πλαίσιο. Να συνειδητοποιήσουμε ένα πράγμα όμω. Ε, οι διατάξει για τη διαρροή άνθρακα απορρέουν από τις, τα συμπεράσματα του Οκτωβρίου 2014 και μα υποχρεώνουν αυτά τα συμπεράσματα να διατηρήσουμε τα ποσοστά σε σχέση με τη δράση των κρατών μελών και από την άλλη πλευρά να μειώσουμε το συνολικό αριθμό αυτών των ε, ε, πιστοποιητικών ώστε να καταλήξουμε σε 1,74%. Τι σημαίνουν και τα δύο λιγότερα πιστοποιητικά για ελεύθερη ε, διάθεση. Αυτό θα σημαίνει ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα τρία, αυτοί οι τρεις άξονες θα υποφελήσουν εκείνους που πιέζονται περισσότερο. Δεν μπορούμε να επιλέγουμε το τι επιθυμούμε σε σχέση με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δεν είναι κάτι το οποίο συμμεριζόμαστε. Το αντίθετο. Πιστεύουμε ότι η συμφωνία που επετέφθη από του ηγέτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση διαφυλάσσει μια πολύ ευαίσθητη ισορροπία, επί τη οποία θα πρέπει να υπάρξει συνένεση αν δεν θέλουμε να υπονομεύσουμε τη συνολική προσέγγιση. Υπό αυτό το πνεύμα και δεδομένου του, του πιο περιορισμένου αριθμού πιστοποιητικών πρέπει να έχουμε μια πιο στοχοθετημένη δράση. Πρώτον, χρειαζόμαστε ένα καλύτερο σύστημα για την επικαιροποίηση των βέλτιστων προδιαγραφών Πρέπει να αντανακλά το σύστημα αυτό των βέλτιστων προδιαγραφών των τεχνολογιών μας ώστε να ανταμείβονται οι πιο επιτυχείς εταιρείε στι επιδόσεις τους και να υπάρχουν κίνητρα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ε, άμεση ευθυγράμμιση σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγή των επιχειρήσεών μας. Αυτό είναι συγκεκριμένο αίτημα των επιχειρήσεων και βιομηχανιών. Τέλο πρέπει να στοχοθετήσουμε καλύτερα του στόχου που, που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερε πιέσει ανταγωνισμού και σε σχέση με τι εκπομπέ τρύπων Πρέπει όμω και το σύστημα να καταστεί πιο δυναμικό και γι' αυτό προτείνουμε να επικαιροποιηθούν τα benchmarks και τα επίπεδα παραγωγή σε τακτά διαστήματα και να εισαχθεί ένα σύστημα με πρόσθετα 400 εκατομμύρια για να υποστηριχθούν οι εταιρείε και εκείνοι που βρίσκονται στην παραγωγή. Χάρη σε αυτά τα στοιχεία οι πιο έντονοι τομείς σε σχέση με την διαρροή άνθρακα θα δουν μια σημαντική μείωση του διατομεακού αυτού ε, στοιχείου αναφοράς. Δηλαδή, αν δεν είχαμε συμπεριλάβει αυτά τα τρία στοιχεία δεν θα υπήρχαν αρκετές άδειε ε, για τον επιμερισμό αυτών των πιστοποιητικών. Θα έπρεπε να υπάρξει μια μείωση συνολικά κατά 35% μέχρι το 2030. Αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, να ολοκληρώσω τι παρατηρήσει μου για την αναθεώρηση του EPS, του συστήματο εμπορία τρύπων. Είναι πολύ σημαντικό για την μείωση του άνθρακα στην ε, ατμόσφαιρα. Η καινοτομία για τι ε, εκπομπέ χαμηλού άνθρακα Θέλουμε να υπάρξει μεγαλύτερη διάθεση κονδυλίων ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις καινοτομία. Θα δημιουργήσουμε ένα ταμείο καινοτομία ώστε να υποστηριχθούν οι τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα και 400 εκατομμύρια θα διατεθούν σε αυτό το ταμείο. 50 εκατομμύρια που ζήτησε το Κοινοβούλιο για αυτό το σκοπό θα προσθεθούν επιπλέον για να ενδυναμωθεί και να καταλήξει σε 450 εκατομμύρια αυτό το ταμείο. Δεύτερον, θα δώσουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη ώστε να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να υποφεληθούν από ένα ταμείο συνοχής νέα λειτουργία για το μέλλον. Και τέλος αυτή η πρόταση απαιτεί μια, ένα πιο εναρμονισμένο και πιο διαφανές σύστημα από πλευρά των κρατών μελών. Ήταν επίσης ένα αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεχτήκαμε. Έτσι οι προτάσει μας καταλήγουν σε μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την δυνατότητα αντισταθμίση. Ε, έχουμε λοιπόν πιο ελαστικού, πιο ευέλικτους και πιο εναρμονισμένου κανόνε. Πιο στοχοθετημένη δράση για τον εξυγχρονισμό του ενεργειακού τομέα. Θα συνεισφέρουμε για την καλύτερη λειτουργία τη ενεργειακή αγορά τη Ευρώπη, ενώ θα ανταποκριθούμε στα αιτήματα των στόχων για μικρότερε εκπομπέ άνθρακα, που θα επιβαρύνουν λιγότερο την ατμόσφαιρα. Πρόκειται λοιπόν για την διάθεση στους ε, καταναλωτές εύληπτων πληροφοριών που θα μπορούν να αντιλαμβάνονται τι, τι συμβαίνει με τα ενεργειακά προϊόντα. Είναι σημαντικό αυτό διότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από εμά προτού αγοράσουν ενημερώνονται σε σχέση με τις ετικέτες και τα στοιχεία. Όλα αυτά θα βοηθήσουν 465 ευρώ να εξοικονομούν οι καταναλωτές ετήσια και θα υπάρξει πολύ μια πολύ μεγάλη συνολική εξοικονόμηση επιπλέον 15, 10 ε, δισεκατομμύρια θα μπορούν να διατεθούν επιπλέον σε επιχειρήσεις και θα εξοικονομηθεί τέτοιο ποσοστό ενέργειας όπως η ετήσια κατανάλωση ενέργειας των βαλτικών κρατών. Αυτό λοιπόν θα μπορεί να είναι μια επιτυχής διαδικασία θα πρέπει να οδηγηθούμε σε διαφορετικά επίπεδα για να μπορέσουμε με τις νέες τεχνολογίες αποτελεσματικότητας να έχουμε κάποια πιο θετικά αποτελέσματα. Από το 2010 όμως τα κινηθήκαμε με ταχύτερους ρυθμούς και ενώ βλέπουμε ότι ε, θεωρούμε ότι ένα προϊόν μπορεί να είναι το πιο αποτελεσματικό στην αγορά, μπορεί να είναι το λιγότερο αποτελεσματικό σήμερα. Έχουν ε, εν τω αλλάξει τα δεδομένα. Προτείνουμε λοιπόν σήμερα να επανέλθουμε σε, ένα, σε μια απλή κλίμακα AG και να έχουμε μια ε, πιστοποίηση των προϊόντων για να μην υπάρξει σύγχυση στη μεταβατική περίοδο και να δώσουμε κίνητρα για τις τεχνολογίες προτείνουμε τρία πράγματα. Τα, κανένα προϊόν δεν θα εισέρχεται στην ε, ε, αλυσίδα ώστε να υπάρξει αυτό το περιθώριο κατά το μέλλον. Δεύτερον, όταν θα έχει σχεδιαστεί ένα τέτοιο προϊόν, η παλαιά ετικέτα θα πάψει να λειτουργεί και θα υπάρξει νέα ετικέτα. Και τρίτον, οι ηλεκτρονικές ετικέτες θα χρησιμοποιούνται ως συμπλήρωμα. Αλλά όλα αυτά θα μπορέσουν να λειτουργήσουν όταν θα αρχίσει η περίοδος λειτουργίας αυτών των ηλεκτρονικών ετικετών και πρέπει να δούμε ότι οι εθνικές αρχές εποπτείας ε, δεν μπορούν να έχουν αυτή την πρόσβαση σε όλες αυτές τις πληροφορίες. Προτείνουμε λοιπόν να υπάρξει μια τράπεζα δεδομένων, ηλεκτρονικού χαρακτήρα, ηλεκτρονική τράπεζα δεδομένων, ώστε να μπορούν οι αρχές εποπτείας των κρατών μελών να δράσουν αποτελεσματικά. Να ενημερώνονται στο τέλος τέλος οι καταναλωτές. Η ενημέρωση χωρίς ε, τις εξουσίες να επιλέγουν όμως δεν έχει νόημα. Η πλατφόρμα δίνει την δυνατότητα να υπάρχει η ε, καθοδήγηση από τους καταναλωτές προς την κατεύθυνση προς την οποία θέλουν να, πρέπει να κινηθούν οι αγορές. Πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη. Μείωση ε, των, τιμών εισαγωγών προϊόντων, μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και να υπάρξει ένα κλίμα το οποίο θα είναι αηφόρο και θα ε, μπορεί να ε, εξυπηρετήσει τις επόμενες γενναίες. <clears throat> αναμένω ότι οι συζητήσεις ε, θα αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις. Μπορούμε όμως αυτές τις προκλήσεις να τι αντιμετωπίσουμε με σκληρή δουλειά και ανοιχτό πνεύμα. Βασίζομαι στην υποστήριξή σας γι' αυτό και προσβλέπω στι απόψεις σας. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον ε, κύριο Επίτροπο για την παρουσίαση τρεις προτάσεις που για μα είναι πολύ σημαντικέ από πλευράς ε, επιτροπής μας είναι εξαιρετικά κρίσιμη σημασία για τα ζητήματα που εμπίπτουν στι αρμοδιότητέ μας, αλλά και για τις μικρομεσαίε επιχειρήσει και για τη βιομηχανία. Τώρα, εξ ονόματο των ε, πολιτικών ομάδων. Από το ΕΛΚΟ, κύριο Κάριντς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τον Επίτροπο. Πολλά είναι τα νέα κείμενα, τα οποία πρέπει να επεξεργαστούμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και βέβαια είναι πολύ καλό που κάνουμε αυτή τη συνεδρίαση. Θα ήθελα να επικεντρωθώ μόνο σε μία πτυχή της ομιλία σας. Πολλά έχω να πω και για τη θύμανση, το ενεργειακό σήμα, αλλά δεν θα επισέλθω σε αυτό. Για τη διακυβέρνηση. Μιλήσατε για το σχέδιο της ενεργειακής αγοράς, το σχεδιασμό. Μία από τις δυσκολίε που έχουμε στο διασυνοριακό εμπόριο είναι ότι αφενό βεβαίω έχουμε και φυσικού περιορισμού. Δεν έχουμε αρκετέ ε, γραμμές μετάδοσης ε, με αρκετή χωρητικότητα για όλα τα κρατημέλη. Άλλο είναι καλύτερα, άλλο είναι χειρότερα. Αλλά εκεί που είναι καλύτερα τα πράγματα, συχνά υπάρχει δυσκολία πρόσβαση ε, στι υποδομέ. Επομένω, ο πάροχο, που δίνει πρόσβαση τα μεσάνυχτα και όχι την ημέρα, ας πούμε, όταν είναι πιο υψηλή η κερδοφορία, αν θέλετε. Πώς προτείνετε να ενισχυθεί ο ρόλος του Acer ε, για, τους, ε, για αρχές ενέργειας, για να γίνουν πιο αποτελεσματικές, από το, τη χονδρική να περάσουμε και στη λιανική και αν λάβει τέτοιο ενισχυμένο ρόλο, πώς αυτό ε, θα συσχετιστεί και με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Είναι σημαντικό να αυξηθεί και να ενισχυθεί ο ρόλος της ρύθμισης στην Ευρώπη για να επιλύσουμε και τέτοια αντισυνοριακά προβλήματα που ξέρουμε ότι και πάλι θα υπάρχουν, ακόμα και αν υπάρχει διασύνδεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά ακριβώς. Τέλεια. Από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Νίκα. Ένα ερώτημα για τα τρία αυτά πακέτα. Κατόπιν της εφαρμογής ε, της υλοποίησής σας θα υπάρξει αύξηση των τιμών της ενέργειας για τον μεμονωμένο καταναλωτή ή και για την βιομηχανία. Και αν ναι, τι τάξη θα είναι αυτή η αύξηση. Πότε θεωρείτε ότι θα υπάρξουν αυτές οι αυξήσεις. Μετά, οι τρεις προτάσεις ακολουθούνται και από μία αξιολόγηση αντικτύπου. Αν υπάρξει τέτοια αξιολόγηση αντικτύπου, θα θέλαμε να το στείλετε αυτό το έγγραφο και στην Επιτροπή μας. Ούτως ώστε αυτά που έχουν συμβεί στο παρελθόν να μην συμβούν και πάλι. Πολλοί συνάδελφοι δεν θέλουν να σας δώσουν μια λευκή επιταγή. Αν υπάρχει αντίκτυπος πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ποιος θα είναι αυτός να είμαστε καταλήλως ενημερωμένοι. Γιατί κάποιοι λένε ότι αυτό το πακέτο, το ETS, θα συζητηθεί μόνο στην ΕΝΒΗ. Μπορούμε να του πούμε όμως ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Πρέπει να ξέρουμε και από πλευρά βιομηχανία σε ποιο θα είναι το κόστο. Και πρέπει να, έχουμε μια... να είμαστε πλήρω ενημερωμένοι για να πάρουμε αυτή την απόφαση. Για να μην ε, υπάρξουν ζητήματα στο μέλλον όπως έχει συμβεί και παλαιότερα. Για την πρόταση για το σήμα, είναι εντελώ νέο το σύστημα. Ποιο θα αναλάβει το κόστο αυτή τη ε, πλήρου αλλαγή του συστήματο, από το Α που είχαμε στο παρελθόν, όταν αγόραζε κανεί ένα ψυγείο, τώρα θα περάσουμε από το A μέχρι και το G. Υπάρχει αξιολόγηση δικτύπου. Ποια είναι η αξιολόγηση δικτύπου, τι λέει. Και σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό της αγοράς, αυτή η μετάβαση από το σύστημα προστασίας του καταναλωτή για τους ευάλωτους καταναλωτές πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά. Αυτή η σταδιακή κατέργηση θα πρέπει να λάβει υπόψη το γεγονό ότι υπάρχει και ενεργειακή ανέχεια. Όπως γνωρίζετε, ε, ο αριθμός αυτών των καταναλωτών είναι πολύ ψηλό στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή και πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Και, κύριε Επιτρόπε, παρακαλώ να μεταφέρετε αυτό το μήνυμα ότι δεν έχει ΑΡ. Δεν μπορεί να το δεχθεί αυτό η ομάδα μας πλέον. Εκτός και αν έχουμε αξιολόγηση αντικτύπου στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ. Εκ ε, του ECR, Μάρικ Γκουβάτσι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Οι νέες προτάσεις που μας μετέφερε ο Επίτροπος προφανώς θα χρειαστεί πολύ καιρό για να τα συζητήσουμε, να τα εξετάσουμε μάλλον σε βάθο. Σε ό,τι αφορά την πρόταση για τη σήμανση και τη μείωση κατανάλωση ενέργεια, είναι κάποιε από τι προτάσει, αλλά οι λύσει που προβάλλονται ε, από ό,τι φαίνεται κινούνται προς μία μάλλον επικίνδυνη κατεύθυνση. Μείωση των εκπομπών επομένω και στις ενεργοβόρες βιομηχανίες, ε, για παράδειγμα στην Χαλιβουργία και στη χημική βιομηχανία. Και εδώ θα είχαμε άμεσο αντίκτυπο στην αγορά σήμανση. Αν θέλουμε να λύσουμε το, τα προβλήματα στην αγορά σήμανση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να εξετάσουμε και τι ενεργοβόρε μα βιομηχανίε. Να τι καταστήσουμε πιο ανταγωνιστικέ. Ακούσαμε λοιπόν αυτέ τι πρώτε προτάσει, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει τρόπο να γίνει αυτό. Δεν νομίζω ότι προσπαθείτε να διασφαλίσετε ότι αυτές οι βιομηχανίες ε, θα φύγουν από την Ευρώπη, εάν είναι κοστοβόρες, ενεργοβόρες μάλλον, συγγνώμη. Ιδίως ότι φορά τη βαριά βιομηχανία. Και με βάση και των προτάσεων για το carbon leakage. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το ζήτημα, αλλά όπως είπα χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να το αναλύσουμε. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο θίξατε, Επίτροπε, αφορά τη μόνιμη ασφάλεια εφοδιασμού. Σήμερα στην Επιτροπή ήδη συζητήσαμε τη νέα συμφωνία μεταξύ Gazprom και ορισμένων ευρωπαϊκών εταιριών στο πλαίσιο του Nord Stream. Και είδαμε ότι σκοπός είναι να αυξηθεί ε, ο εφοδιασμός, η παροχή φυσικού αερίου, να διπλασιαστεί σχεδόν στα 100 δις ε, κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην Ευρώπη που θα παρέχονται από την Gazprom. Ποια είναι η θέση σας και πώς σας σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε αυτό το ότι μάλλον επικίνδυνη συμφωνία κατά τη γνώμη μου. Έχουμε αυτερικές επιχειρήσεις, την άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες. Πώς θα το αντιμετωπίσετε. Ο κύριο Φέντριλε, εκ μέρου τη Άλντε. Ευχαριστώ πολύ Προέδρε, ευχαριστώ για να και σας κύριε Επίτροπε. Η Επιτροπή μα έχει πολύ σημαντικό καθήκον εδώ. Την περασμένη φορά είχαμε το MSR επιτάπητο και αποτύχαμε πλήρω. Καταψηφίστηκε η ε, γνωμοδότηση και αυτό δεν είναι προ όφελο τη βιομηχανία μα. Και εμεί έχουμε τη δική μα προοπτική και οπτική γωνία αν δεν έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα, το αυτό αποτελεί αποτυχία. Αν ζητούμε τη δικασία του άρθρου 55, τότε πρέπει να έχουμε και ε, τα απαραίτητα αποτελέσματα. Είναι σημαντική ευθύνη λοιπόν για μας. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το σημείο εστίασης να είναι οι Θα είναι θετική αλλαγή. Σίγουρα ένα σημείο προόδου. Είμαι υπέρ του Ταμείου Καινοτομία. Καλό είναι να κλείσει, να περιοριστεί ο κατάλογο του carbon leakage, ιδίω για την ευρωπαϊκή βιομηχανία σημαντική είναι η αναθεώρηση του σήματο, που νομίζω ότι έχει αποτελέσει πρόβλημα για τη βιομηχανία. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά όμως τις επιπλέον ε, ελεύθερες άδειες ε, και πιστοποιητικά για την Ανατολική Ευρώπη, βελτιώνει, ενισχύει μάλλον τη στρέβλωση στην ηλεκτρική ενέργεια, το είπαμε και σήμερα το πρωί. Γιατί δίνουμε χαμηλότερε ε, τιμέ ενέργεια σε κάποια τμήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και υψηλότερε τιμέ αλλού. Η Πολωνία, για παράδειγμα, θα έχει πολύ μεγάλο όγκο και αριθμό δωρεάν πιστοποιητικών που θα ρίξει τις τιμέ στην Πολωνία της ηλεκτρικής ενέργειας, όχι επειδή έχουν όμως ε, εύρυθμη λειτουργία της αγοράς που οδηγεί σε χαμηλέ τιμέ και θα αυξήσει ε, τις ε, τιμές στο βορρά. Δεύτερον, το επίπεδο φιλοδοξία. Θα μπορούσε να είναι και ανώτερο και θα τυχεία. Με προβληματίζει λίγο το πώς τα έσοδα αυτά που θα προκύπτουν από τις δημοπρασίες αξιοποιούνται στα κράτη-μέλη γιατί αυτά τα χρήματα υποτίθεται ότι θα δίνονταν ε, στο δρόμο των απαλλαγμένων από άνθρακα. Αλλά συμβαίνει αυτό. Στη Σουηδία, για παράδειγμα, εμείς ε, πουλήσαμε αυτές τις ε, άδειε και τις αξιοποιήσαμε για να πληρώσουμε το δημόσιο χρέος. Αυτό κάναμε λοιπόν. Πρέπει λοιπόν να αξιοποιούνται αυτά τα χρήματα ακριβώ για το σκοπό που είχαμε ω στόχο. Μετά, αποζημίωση ό,τι αφορά τι δευτερογενέ επιπτώσει στην ηλεκτρική ενέργεια. Πρέπει η αποζημίωση να την χάνει η ίδια μεταχείριση σε, σε επιμέρου κρατημέλη. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, το 100% προκύπτει από, από το δημόσιο, ενώ αλλού δεν υπάρχει καμία αποζημίωση. Και έτσι υπάρχει στρέβλωση και πάλι στην εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Αρχικά έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο ότι πρέπει να υπάρξει μεταρρύθμιση και εμεί θέλουμε να, να επανέλθουμε στο A2G, όχι στο A++ πλέον. Δεύτερον, το πακέτο σας για το σχεδιασμό της αγοράς είναι πολύ καλά καταρτισμένο. Λέτε ότι ο καταναλωτής πρέπει να μπει μπροστά. Είναι μια καλή προσέγγιση. Με τις νέες τεχνολογίες μπορούμε να δώσουμε μεγαλύτερο ρόλο στους καταναλωτές. Και ο σχεδιασμός της αγοράς, αυτό το έγγραφο είναι πολύ καλό. Ε, προετοιμάζει την αγορά για τις ΑΠΕ, μιλά για την ηλιακή ε, και ολική ενέργεια, περισσότερη ε, ισχύ στον Acer και μεγαλύτερη ολοκλήρωση σε μακροπεριφερειακό επίπεδο. Ακριβώς αυτό πρέπει να κάνουμε για να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας. Και για πρώτη φορά νομίζω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζεται ότι το πρόβλημά μας είναι η υπερβολική χωρητικότητα και όχι η έλλειψη αυτής σε συγκεκριμένο σημείο αναλύεται πολύ καλά ότι υπάρχει αυτό το overcapacity. Μόνο ένα στοιχείο λείπει από το σχεδιασμό της αγοράς που είναι το εξής. Όταν εγώ βάζω PV στην οροφή μου πρέπει να ε, είμαι συνυπεύθυνος. ακόμα και όταν στο τέλος θέλω να το απομακρύνω από την οροφή μου. Πρέπει λοιπόν να τεθούν κατά μέρος 700 εκατομμύρια ε, για όταν θα έρθει η στιγμή να παροπλιστούν. Αυτές είναι υποχρεώσεις για τις ΑΠΕ, σε ό,τι αφορά λοιπόν ε, την απομάκρυνση αυτών των στοιχείων. Στο πυρηνικό εργοστάσιο δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη. Το διπλάσιο του ελληνικού χρέους, 500 δις, λείπουν ξαφνικά γιατί δεν υπάρχουν ε, ε, χρήματα για την διαχείριση των αποβλήτων. Η Κομισιόν υποσχέθηκε το 2004 ε, να το αντιμετωπίσει και ο Επίτροπος Έτιγκερ με τη Φουκουσίμα είπε ότι εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε όπως έγινε, αυτά που κάναμε με την ΤΑΠΚΟ. Η ΤΑΠΚΟ πτώχευσε και οι Ιάπωνες είναι αυτοί που πληρώνουν την ύφη για μια ζημιά δισεκατομμυρίων. Επομένως, εμείς τι κάνουμε σε μια αγορά που ένα τμήμα της βιομηχανίας και μάλλον η Επιτροπή είναι εντελώς τυφλή. Ακόμα μισό λεπτό δώστε μου, Πρόεδρε, για το ETS. Και ο Φρέντρικ τον ανέφερε. Δώσατε αυτό το δώρο στην ε, Πολωνία, στην PGE, για τις ελεύθερες αυτές δωρεάν άδειες. 30 δις για μια χούφτα Επιχειρήσει. Αντί να τις δημοπρατήσετε αυτές τις άδειε και οι Πολωνοί να ανακαινήσουν τα κτίρια τους. Ουσιαστικά η Πολωνία έχει υψηλότερες τιμές ενέργειας από ό,τι στη Γερμανία ή από ό,τι στη Σκανδιναβία. Υπάρχει λοιπόν τέτοια διαρροή από την Πολωνία, όχι όμως προς τη ΣΥΠΑ, αλλά προς τη Γερμανία και προς τη Σκανδιναβία γιατί αυτές οι χώρες μαζί με τη Γαλλία έχουν χαμηλότερες τιμές επειδή υπάρχει και διασύνδεση. Παρακαλώ εξετάστε την πραγματικότητα ε, πίσω από αυτό το δώρο των 30 δις. Από την ΚΟΕ, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ο, ο σχεδιασμός της αγοράς του ηλεκτρικού είπαμε πολλές φορές πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο τις να έχει στο επικέντρο της ανάγκης της κοινωνίας. Χαιρόμαστε γιατί τίθεται το θέμα ότι πρέπει στο επικέντρο να είναι ο καταναλωτής. Πρωταρχικός στόχος για, για αυτό είναι να διασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια σε ηλεκτρικό ρεύμα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να αρθεί η ενεργειακή απόμονωση κρατών και περιοχών από τα μεγάλα ηλεκτρικά δίκτυα. Δηλαδή είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι ελληπείς υποδομές και να προωθούν νέε ολοκληρωμένε προτάσει ώστε να επιτύχουν όλε οι χώρε το στόχο που έχει τεχθεί για το 10% τη ηλεκτρική διασύνδεση ω το 2020. Είναι βεβαίω ε, αναγκαίο και σημαντικό να προωθούν μέτρα για καταπολέμηση τη ενεργειακή φτώχεια και μείωση του κόστου του ηλεκτρισμού, ηλεκτρικού ρεύματο, ιδιαίτερα για του καταναλωτέ, τα νοικοκυριά, ε, του μικρού παραγωγού και τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, ε, ένα σύστημα που εφαρμόζεται σε κάποιες χώρες, το γνωρίζω γιατί ε, το έχω ξεκινήσει ως πιλωτικό πρόγραμμα όταν ήμουν Υπουργός Ενέργειας στην Κύπρο, είναι το σύστημα του net metering, του ηλεκτρικού συμψηφισμού, δηλαδή με τη χρήση ανανόσιμων πηγών ενέργειας. Ένα σύστημα που βοηθά πάρα πολύ τα νοικοκυριά ε, σε αυτήν την κατεύθυνση για να έχουν φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα αλλά ταυτόχρονα αυξάνουμε και τη συμμετοχή των, α, των ΑΠΕ και θα ήθελα να ρωτήσω εάν ε, σχεδιάζουμε κάποια μέτρα ε, σε αυτή την κατάσταση ε, για να μπορέσουμε να ελαφρύνουμε τα νοικοκυριά. επίσης κύριε Επίτροπε, στις εκτιμήσεις της Επιτροπής είναι ότι υπάρχουν ενεργειακά απομενωμένα κράτη τα οποία δεν μπορούν να υλοποιήσουν αυτό το στόχο όπως είναι η Κύπρος. Ένα θετικό βήμα για λύση του προβλήματος είναι να προχωρήσει ένα έργο ε, το γνωστό ε, Euroasian Interconnector είναι η διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδα, το οποίο έχει ενταχθεί στα έργα κοινού ενδιαφέροντο. Ε, η ολοκλήρωση του έργου αυτού σε συνδυασμό με τι ενεργειακέ πηγέ θα βοηθήσει ακριβώ το ένα από τη μια να, να διοχετευτεί φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, αλλά να έρθει και η απομόνωση ενό κράτου μέλου όπω είναι Κύπρο και ήθελα να ρωτήσω πώ θα προωθήσει ε, αυτών τον έργο πώς θα το στηρίξει η Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you very much, colleague. Ευχαριστώ κυρία Κάπελ από το ΙΕΝΕΦ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε Κανιέτα για την παρουσία, παρουσίαση του θερινού, της θερινής δέσμης μέτρων summer packages και ότι λάβατε υπόψη και το New, το New Deal, τη νέα συμφωνία τα στοιχεία που προτάθηκαν είναι πολύ σημαντικό. Πρόκειται πραγματικά για τη διαμόρφωση προσιτών τιμών, πιο χαμηλών τιμών για τους καταναλωτές, αλλά και με τις νέες τεχνολογίες που θα εισαχθούν, ψηφιακές τεχνολογίες και ένα μέσο για τις αγορές, ώστε είναι αξιοχαιρέτιστο το ότι πραγματικά θα μπορέσουμε να κινηθούμε ώστε μέτρα της αγοράς να μπορέσουν να προαθούν υπέρ των καταναλωτών. Πολύ θετικό βήμα. Σημαντικός είναι και ο σχεδιασμός της ηλεκτρικής αγοράς ε, design και είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη και τα συστήματα όσον αφορά τις διαδικασίες ε, αντιμετώπισης των στρεβλώσεων ε, πέρα από τα, τα σύνορα των κρατών μελών και να λάβουμε υπόψη και το δυναμικό των αγορών. Είπατε ότι δυναμικές αγορές ή η διαμόρφωση τέτοιων αγορών θα πρέπει να οδηγήσει και σας ερωτώ πώς θα διασφαλίσετε αυτούς τους στόχους που παρουσιάσατε. Λέτε επίσης ε, ότι θα μεριμνάτε για τις ε, διασυνοριακές ροές ε, ενεργειακών προϊόντων. Στην Αυστρία οδηγούμαστε στο ότι η ζώνη αυστρογερμανική για τις ενεργειακές τιμές αφορά και τα θέματα της διασύνδεσης και θα πρέπει έτσι να εξετάζεται. Ερώτησή μου, κινείστε με προς μια ενιαία κατεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την ενεργειακή ζώνη τιμών Γερμανίας-Αυστρίας και τι θα γίνει δεδομένης της αντιμετώπισης ή κατάργησης αυτής και πώς είναι δυνατόν να υπάρξει ε, τέτοια ρύθμιση με βάση αυτές τις ε, γραμμές ή αν καταργηθούν τι θα γίνει σε σχέση με τις βέλτιστες πρακτικές Επιτρέψτε μου κάποιες παρατηρήσεις για τη μεταρρύθμιση, την αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας ρήπων. Αναφερθήκατε, εγκρίθηκε στο Στρασβούργο το αποθεματικό αγοράς. Ερωτώ τι θα γίνει με την διαρροή άνθρακα. Θέλετε 2,2% ετήσια να υπάρξει μείωση ανά σε σχέση με τα πιστοποιητικά. Πόσο επρόκειται αυτή τη δράση μέχρι το 2020 να την οδηγήσετε στο 20%. Πώς θα το διασφαλίσετε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά από τις πολιτικές ομάδες. Και τώρα θα ήθελα να δώσουμε το λόγο και πάλι στον κύριο Επίτροπο για να απαντήσει. Πρώτα απ' όλα, μία πρώτη παρατήρηση γενική. Όταν προετοιμάσαμε την ε, πρόταση για το ETS κατά βάση, λάβαμε την απόφαση να παρακολουθήσουμε εκ των στα και να ακολουθήσουμε μάλλον τα αποτελέσματα του, Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου του 2014. Ήταν σημαντικό να υπάρχει μια ισορροπία, γιατί όλοι ε, δέχονταν ε, τους φιλόδοξους και ισορροπημένους αυτούς στόχους είναι μια σορπημένη λοιπόν συμφωνία και έτσι αποφασίσαμε όσο Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μείνουμε εκεί. Να κάνουμε μια πρόταση κατά το δυνατόν καλύτερα καταρτισμένη, αλλά με βάση αυτό το πακέτο. Και το πακέτο που είναι το κύριο στοιχείο υπήρχε σαφής ένδειξη ότι η κατανομή των ε, αδειών μεταξύ της δημοπρασίας και των δωρεάν αδειών προς τη βιομηχανία δεν πρέπει να αλλάξει. Και αυτός ο κατάλογος με τους 57 για τη δημοπρασία και οι υπόλοιπους για τη βιομηχανία. Αυτό είναι το σημείο κίνησης. Δεν μετακινηθήκαμε από εκεί. Και το δεύτερο είναι ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επίσης αποφάσισε ότι για να υπάρξει αυτή η μείωση κατά 43% στο ETS γιατί στην τομέα του ETS δεν είναι 40% της μείωσης, είναι 43%. Ο αριθμός των ε, αδειών πρέπει να μειώνεται κάθε χρόνο κατά 2,2%. Δεν έχω εδώ τα στοιχεία μου. Κάπου τα είχα, αλλά πάντα τα χάνω. 500 ή μάλλον 48 εκατομμύρια κάθε χρόνο θα μειώνονται κάθε χρόνο λοιπόν οι άδειε. Στην περίοδο έως 2030 μετά θα υπάρξει μείωση 536 εκατομμυρίων αδειών. Υπάρχει λοιπόν σημαντική προσπάθεια μείωση των εκπομπών και μισό εκατομμύριο, μισό δις λιγότερες άδειες. Πρέπει να λύσουμε το ζήτημα του carbon leakage. Πρέπει να γίνει μια δίκαιη και ισόρροπη ε, πρόταση που είναι εξαιρετικά δύσκολο, όπως σας λέω, γιατί με αυτά τα στοιχεία αν είχαμε μείνει στην πεπατημένη, κάθε βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είχαν μείωση 35% με έναν συντελεστή διόρθωση, αν δεν είχαμε κάνει τίποτα. Εμείς τι κάναμε τώρα για να διαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα που να στοχεύει περισσότερο αυτούς που πρέπει να αφαιρέσουμε τον συντελεστή διόρθωση αυτό ε, κατά το δυνατόν. Είναι λοιπόν μία πολύ ε, επεξεργασμένη, αν θέλετε, πρόταση και ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Με την πλήρη συνεργασία του επιτελείου μου, των συναδέλφων μου, για να δώσουμε όσο γίνεται περισσότερες πληροφορίες. Θα έρθω με την ε, αξιολόγηση που Θα τη δώσω σε όλα τα μέλη της Επιτροπή. Δεν κρύβουμε τίποτα εδώ πέρα. Να ξέρετε και τις δυσκολίε. Γιατί αν αγγίξουμε και μετακινήσουμε ένα κομμάτι του πάζελ, μετακινούνται και τα υπόλοιπα. Δεν είναι ασύνδετο. Αυτό είναι μια πρώτη παρατήρηση. Θέλω να συμμετέχω, να συμμετέχω πλήρως στην Επιτροπή σας για να τα εξηγήσω όλα, εμεί είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε πρόταση, όμω σα διαβεβαιώ ότι αφιερώσαμε πολύ χρόνο για να ε, προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε έναν μηχανισμό υπό το ευρύτερο πλαίσιο που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αν αλλάξουμε το πλαίσιο θα αλλάξει και η πρόταση. Αν όμως στηρίσουμε το πλαίσιο που ήταν ε, μία λεπτή συμφωνία και τελευταία στιγμή και ο πρόεδρος ε, τη Επιτροπή το γνωρίζει πόσο δύσκολη ήταν αυτή η συμφωνία. Είναι λοιπόν... Ε, ε, βεβαίω, τώρα για να απαντήσω, πράγματι υπάρχει πρόβλημα με τη συνεργασία των PSOs. Γιατί πράγματι χρειαζόμαστε υποδομέ, διασύνδεση για να έχουμε του στόχου αυτού του 10 και 15%. Θέλουμε διασύνδεση και στο φυσικό αέριο, αλλά πρέπει να ενισχύσουμε ε, τη συνεργασία μα. Ιδάλω δεν θα έχουμε πραγματικά ευρωπαϊκό δίκτυο. Υπάρχουν πολλέ πρωτοβουλίε εθελοντική ε, περιφερειακή συνεργασία και έχουμε και συγκεκριμένο ε, σύστημα που θα ψηφιστεί στην Επιτροπολογία στη συνέχεια της χρονιάς και θα προτείνουμε την δημιουργία των πρωτοβουλειών συντονισμού, περιφερειακού συντονισμού σε όλη την Ήπειρο. Σημαντικό βήμα για περαιτέρω περιφερειακό συντονισμό και συνεργασία για την διαχείριση συστημάτων. Ιδάλλως δεν μπορούμε να ενσωματώσουμε και τις ΑΠΕ στο δίκτυο. Πρέπει να γίνει λοιπόν αυτό. Και επίσης η συμβουλευτική ανακοίνωση σε αυτή την πρωτοβουλία για το market design θα εξηγήσει πώς θα βελτιώσουμε αυτή την πρωτοβουλία. Θα επανέλθουμε λοιπόν με νομοθετικέ προτάσεις του χρόνου για να λύσουμε αυτό το ζήτημα. Μετά έχουμε το στήμα του Acer. Είναι σαφέ. για μια εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, ο Acer θα διαματήσει πολύ σημαντικό ρόλο. Και ο Acer πρέπει να παρακολουθεί τις ε, αγορές χοντρική για να αποκαλύπτει στρεβλώσεις και καταχρήσει ε, στην αγορά Απαιτούνται πόροι, εμπειρογνωμοσύνη, γι' αυτό και εμείς προτείναμε να αυξήσουμε το προσωπικό του Acer στον προπολογισμό του 2016, θα δούμε αν θα το επιτύχουμε. οι συνομοθέτες θα το αποφασίσουν, όμως θέλουμε να εφαρμόσουμε τις αρμοδιότητες του Acer. Θα δούμε και τις ε, απόψεις του Κοινοβουλίου. Βεβαίω θα σα δώσουμε τι αξιολόγηση αντικτύπου, όπω είπα και προηγουμένω, προ τον κύριο Νίκα. Η αξιολόγηση αντικτύπου είναι κάτι που παίρνουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Ήταν δύσκολο για την πρόταση ETS να περάσει η αξιολόγηση αντικτύπου. Υπήρξαν προβλήματα στην αρχή. Έπρεπε να κάνουμε και περαιτέρω εξηγήσει και διευκρινήσει, όμω θα δείτε όλα τα δεδομένα και στοιχεία. η κατανάλωση είναι εξαιρετικά σημαντική και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε γιατί αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο να έχουμε κοινή προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα τα κράτη-μέλη κάνουν ο καθένα το δικό του. Κάποιοι απαγορεύουν, την, μάλλον την αυτόνομη παραγωγή. Ε, άλλοι το απαγορεύουν, άλλοι το φορολογούν. Πρέπει να έχουμε λοιπόν τουλάχιστον περιφερειακές ε, λύσεις ω προς αυτό. Κύριε Γκρομπάτσκι, για την χημική βιομηχανία και το carbon leakage. Η χημική βιομηχανία θα είναι από τις, ε, τους 50 κλάδους που έχουν 100% δωρεάν άδειε. Είναι ενεργοβόρες, γιατί στο σχεδιασμό αυτών των ε, τομέων συνδυάζουμε την ένταση ενέργειας με άλλα στοιχεία. Η Κομισιόν έχει σαφείς απόψεις. Από πλευράς ε, ασφάλειας εφοδιασμού, το σημαντικό για μας είναι ο νότιος διάδρομος. Η διασύνδεση με το Αζερβαϊτζάν, εναλλακτική παροχή σε σχέση με τη Ρωσία, Τουρκμανιστάν, Ιράν. Στο μέλλον, ίσως μπορεί να έχουμε και διασύνδεση με το δίκτυο του Ιράν. Και έτσι θα υπάρχει διαφοροποίηση. Για τον Nord τα πράγματα είναι διαφορετικά ο ιδιωτικό τομέα ε, καταλήξει στη συμφωνία και λέει ότι θέλει να στήσει νέον φυσικό αγωγό. Η θέση τη Επιτροπή είναι σαφή. Εμεί θέλουμε το φυσικό αέριο να περάσει από την Ουκρανία. Δεν πρέπει να παρακαμφθεί. Και αν θέλουν τον Nord Stream, που δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, τότε θα πρέπει να συμμορφωθούν με το τρίτο πακέτο ενέργεια, με του κανονισμού δημοσίων προμηθειών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μας προτεραιότητα είναι η διαφοροποίηση των παρόχων. Να υποστηρίξουμε τον νότιο διάδρομο. Πήγαμε και στην Κροατία. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Έχουμε δική μας στρατηγική. Με την Gazprom και τους υπολείπους. Εμείς, εμάς μας νοιάζει η ασφάλεια εφοδιασμού. Κύριε Φέντερλε. Κάνοντας λόγο για το ταμείο αυτό, αυτό δεν αναφέρεται. Και αν οι στρεβλώσεις ε, που θα δημιουργούνται στις αγορές ε, θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν 2% των 57% όσον αφορά τις ε, τους πληστηριασμούς και θα είχαμε 10 εκατομμύρια που θα οδηγούσαν στην, συνολική αξία 7 δις ευρώ και θα διασφαλίζαμε να ότι θα χρησιμοποιηθεί αυτό το ποσό σύμφωνα με τις αρχές που εμπνέουν το σύστημα εμπορίας ρήπων ETS και φυσικά το ταμείο αυτό δημιουργήθηκε με τη συμφωνία του Οκτωβρίου και υπάρχει και πρέπει να συμμορφωθούμε με τις διατάξεις του. Κύριε Τούρμες, στην παρέμβασή σας επικεντρωθήκατε σε μία πτυχή που απουσιάζει όσον αφορά τις προτάσεις της Επιτροπής, ιδιαίτερα όσον αφορά και τα πυρηνικά. Θα επανέλθουμε σύντομα με το PINC τη δυνατότητα δηλαδή επικέντρωσης στις επενδύσεις για τους πυρηνικούς αντιδραστήρες και από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ξεκινήσουμε με τις προτάσεις μας πώς θα πρέπει αυτό το πρόβλημα μελλοντικά να αντιμετωπίζεται. Επίσης, ένα θέμα πλεονάσματος δυναμικού αναφέρατε ότι υφίσταται. Είναι σαφές το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν έχουμε την επάρκεια της δημιουργίας, της παραγωγής δυναμικού. Αν το δείτε στο διεθνές επίπεδο, ίσως μπορεί να υπάρξει μια λύση. Αλλά πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση του δυναμικού γενεών σε ένα διαφορετικό επίπεδο και αυτό δημιουργεί ίσως διαφορετικά δεδομένα θα πρέπει να δούμε τα διάφορα δυναμικά και τότε μπορεί κανείς ε, διαφορετικά συμπεράσματα να συναγάγει. Πρέπει να δούμε, θα ενταχθούν τα ανανεώσιμα και ποιες επιπτώσεις θα υπάρχουν. Έχουμε μια σαφή διαδικασία διαβούλευσης που προβλέπεται με στοχοθετημένα ζητήματα που πρέπει να ε, ε, ευθυγραμμίζονται με αυτά οι εμπλεκόμενοι Πρέπει όμως να δούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πλεονάζον δυναμικό επειδή κυρίως ε, η ένταξη των ανανεώσιμων ε, σε σχέση με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα έχουμε 50% της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται από τα ανανεώσιμα το 2030. Θα έχουμε λοιπόν ε, σε σχέση με τα πυρηνικά και την απάλληψη της γενεάς των ορυκτών καυσίμων αλλά 50% της ηλεκτρικής ενέργειας θα παράγεται τότε από τα ανανεώσιμα. Είναι ένας στόχος που έχει εξεταστεί και πρέπει να ενταχθούν τα ανανεώσιμα σε αυτή την πολιτική ώστε να υπάρξει η δυνατότητα υποστήριξης και διασφάλισης νομικής backup ώστε σε σχέση με την παραγωγή αυτή να γνωρίζουμε τι θα γίνεται με, τις, ε, με την κάλυψη των δαπανών και να ξέρουμε σε σχέση με 11 ευρωπαϊκά κράτη ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Θα αναμείνουμε τα αποτελέσματα αυτή τη έρευνα προτού υποβληθούν κάποιες, ε, κάποια μέτρα για την ε, κάλυψη των δαπανών. Αν χρειάζεται κάτι τέτοιο θα πρέπει να δούμε σε ευρωπαϊκό ή περιφερειακό επίπεδο πώς θα διαμορφωθεί και τι θα γίνει με την επανακατανομή σε σχέση με τις, η ε, δυνατότητα ανακατανομής θα ε, προέρθει από τη Συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται σε σχέση με το 10β ή το 10γ ε, για το Ταμείο Εξυγχρονισμού θα υπάρχουν τα κονδύλια του Ταμείου Εξυγχρονισμού και θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις πολιτικές αποφάσεις που θα έχουν ληφθεί και θα ισχύουν. Έτσι λοιπόν θα ανταποκρίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις τοποθετήσεις του Συμβουλίου και όταν θα προτείνει κάτι το Ευρωκοινοβούλιο θα τοποθετηθεί αντίστοιχα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από αυτού. Έχουμε όπως είπα προηγούμενα κάθε σεβασμό σε σχέση με αυτή την πολιτική στοχοθέτηση. Φοβούμαστε ότι αν διαδείξουμε αυτό τον ευαίσθητο πολιτικό συμβιβασμό όσον αφορά τις ισορροπίες των διαφορετικών στοιχείων θα υπάρξει ζημιά. Ακολουθήσαμε λοιπόν την πιο συνετή προσέγγιση. Ο κύριος Σιλικιώτης έκανε λόγο για την ενεργειακή φτώχεια και είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί 11% των ε, ε, πόλεων στην Ευρώπη των νοικοκυριών αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα και πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα της ενεργειακής φτώχειας. Θα εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Και υπό το φόρουμ του Λονδίνου εξετάζονται οι καλύτερες δυνατότητες ή σε σχέση με το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματο ή με την κοινωνική πολιτική των κρατών μελών ή με την πολιτική καλύτερη αποδοτικότητα ενέργεια από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δούμε πώ θα διαμορφωθούν αυτά μελλοντικά, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το μεγάλο, το μείζον πρόβλημα τη ενεργειακή φτώχεια. Η κυρία Κάπελ έκανε λόγο για μηχανισμούς δυναμικού επίσης και για την ε, ε, ανάπτυξη των ε, μικρών αυτών μετρητών όσον αφορά τους καταναλωτές για την διαμόρφωση, δυναμική διαμόρφωση τιμών. Σε βόρειες χώρες έχει οδηγήσει αυτό σε μείωση του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές σε πάνω από 30%. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο αποτελεί θετική επίπτωση αυτού του μηχανισμού. Και όσον αφορά και τον, ε, τις δυνατότητες των μηχανισμών δυναμικού, είπα ότι η επάρκεια της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο και να αξιολογείται σε περιφερειακό επίπεδο προτού θεσπιστούν τέτοιοι μηχανισμοί δυναμικού. Αυτά είχα να πω πρόεδρε για τις παρεμβάσεις ε, και στη συνέχεια μπορούν να υπάρξουν κάποιες πρόσθετες ε, συμπληρώσεις, παρατηρήσεις κτλ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Έχουμε 7 εγγεγραμμένα μέλη στον κατάλογο. Θα ήθελα να σας ζητήσω από ένα λεπτό ο καθένας. Κλείνω τον κατάλογο, ζητώ συγγνώμη. Εντάξει, 30 δευτερόλεπτα ο καθένας σας, ε, συνάδελφοι. Μα κοιτάξτε, ζητώ συγγνώμη, Εντουάρ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε... Όχι, σταματάει ο κύριος Μαρτά. Ωραία, έχω εννέα εγγεγραμμένους συναδέλφους από ένα λεπτό ο καθένας και μετά θα έχουμε την απάντηση ε, του κυρίου Επιτρόπου και θα αρχίσουμε μετά με καθυστέρηση την ε, την ε, συνεδρίαση των συντονιστών. Δεν είσαι ικανοποιημένο, Εντουάρ, από ό,τι βλέπω, ε. Η κυρία Γκρίφιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ, Επίτροπε συλλογικά θα πρέπει να δουλέψουμε έτσι ώστε να ξεριζώσουμε ε, την ε, ενεργειακή φτώχεια. Μια συγκεκριμένη ερώτηση. Έρευνα, πρόσφατη έρευνα αγοράς ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο από την αρχή ανταγωνισμού και αγοράς συμπεραίνει ότι υπάρχει υπερχρέωση της ενέργειας. Ε, γι' αυτό λοιπόν καλωσορίζω αυτή τη νέα συμφωνία New Deal για τους καταναλωτές. Ε, με τον τρόπο αυτό θα γίνει πιο ε, οικονομικά προσιτή η ενέργεια. Και βεβαίως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλοι οι παίκτες και οι φορείς. Υπάρχει βέβαια μία αντίφαση. Η Ενεργειακή Ένωση προωθεί ε, ένα προχωρημένο σχέδιο ενεργειακού συστήματος, ενώ από την άλλη πλευρά ε, ε, προωθούμε και την, αυτο, την αυτάρκεια και την αυτοπρομήθεια. Το αναφέρατε λίγο, μπορείτε να πείτε δυο λόγια παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κάλλας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε που ήρθατε για να μιλήσετε για τα θέματα αυτά. Ο σχεδιασμός της ηλεκτρικής αγοράς είναι πραγματικά κάτι σημαντικό. Μ' αρέσει εκεί που λέει το δανακοινοθένα ότι ε, θα πρέπει να ε, βράχει πρόθεσμα να σχεδιαστεί η αγορά έχοντας κατά νου τις μελλοντικές ανάγκες. Άρα εδώ βλέπουμε και τη διασύνδεση ανάμεσα σε λιανική και χονδρική ε, με τρόπο ώστε εν τέλει να ωφεληθεί ο καταναλωτής. Ένα ζητούμενο βεβαίως εδώ είναι η διαφάνεια και βλέπουμε αυτό που μας ενδιαφέρει ιδιαιτέρωση είναι να υπάρχει συλλογή δεδομένων ε, και συγκριτική ε, αναφορά τους έτσι ώστε να ξέρουν ε, καθαρά οι καταναλωτές πού μπορούν να προμηθευτούν φτηνότερη ενέργεια. Τελευταίον, capacity mechanism. Εάν αναπτυχθούν σε εθνικό επίπεδο, τότε έρχεται σε αντίθεση με την έννοια της Ενεργειακής Ένωσης. Εμείς θέλουμε ε, διασυνδεδεμένη αγορά. Αυτό σημαίνει ότι ε, ίσως θα πρέπει να λειτουργήσει αυτό σε πολλά επίπεδα και σε πολλές ε, χώρες. Ποια είναι η ευρωπαϊκή προσέγγιση, η άποψή σας για αυτό το capacity mechanism, πρόεδρος. Συνάδελφοι, τον Σεπτέμβρη θα καλέσουμε τον Επίτροπο για να συνεχίσουμε την ίδια συζήτηση. Είναι απολύτως απαραίτητο κάτι τέτοιο, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω πράγματι δεν έχουμε χρόνο για ευρεία και σε βάθος συζήτηση. Συμφωνεί ήδη ο Επίτροπος. Το Σεπτέμβρη λοιπόν θα έχουμε τότε το Σεπτέμβριο συζήτηση σε βάθος. Έχω ακόμα έξι συναδέλφους από, έναν, από ένα λεπτό ο καθένας. Ο κύριος Μαρτάν. Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι ε, δικό μου πρόβλημα, δηλαδή δεν ευθύνομαι εγώ για την καθυστέρηση. Κύριε Επίτροπε, έκανα έκθεση για την βιομηχανία. Πήγα σε 8 χώρες, μεταξύ των οποίων ε, και την Ισπανία και πέρα από, την, ε, το κόστος της ενέργειας ε, παραπονιούνται οι φορείς ε, για την έλλειψη προβλεψιμότητας. Αυτή, τι θα κάνετε γι' αυτό, γιατί μιλάμε συνέχεια για χαμηλές ανθρακούγες εκπομπές, αλλά σταθερότητα δεν υπάρχει. Δεύτερον, ε, διαπιστώνουμε ότι ε, έχουμε πρόβλημα όσον αφορά τις επενδύσεις. Το, το κέρδος είναι πάρα πολύ χαμηλό και επομένως ε, δεν ενθαρρύνονται οι, προ, οι επενδύσεις. Τρίτον, μέτρα τα οποία μπορεί να φαίνονται προστατευτικά ε, και, και μέτρα προστατευτισμού, αλλά στην ουσία απλώς φέρνουν μια ισορροπία στην αγορά. Δεν είναι δυνατόν ε, να μην... Ε, Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Μόλις σε μία από τις πιο μικρές ομάδες δώσατε τέσσερα λεπτά και εγώ πρέπει να περιοριστώ τώρα, δεν νομίζω να είναι δίκαιο. Τώρα, μια και είμαστε σε ποσοστώσεις και κάνουμε λόγο για ποσοστώσεις, φυσικά πρόσεξα ότι ο κύριος Κανιέτε στο έγγραφό του για τον λόγο που εξεφώνησε για τον τομέα εκείνον περί του οποίου γίνεται λόγος, ίσως 5 ή 10% έκανε λόγο για το κόστος, την ανταγωνιστικότητα, για την πληττόμενη βιομηχανία. Τα υπόλοιπα ήταν κανονισμοί, διατάξεις, ρυθμίσεις. Ας το πω έτσι, στην Επιτροπή Βιομηχανίας δεν έχουν σωστή κατανομή των βαρών αυτές οι προτάσεις στο τέλος τέλος ε, θα πρέπει να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τις ε, προτάσεις που μας παρουσιάσατε. Αυτή είναι μια συμβουλή που έχει καλές προθέσεις. Τώρα, όσον αφορά την εποπτεία και την παρακολούθηση, θα υπάρξει νέα ετικετοποίηση και λέω με μια ψηφιακή τράπεζα λέει δεδομένων και εποπτεία της αγοράς και ταυτόχρονα θα υπάρξουν ε, εκπομπές ρήπων με τηλεανάλυση. Όλα αυτά είναι πράγματα που με τρομάζουν Κάποτε θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα δίνουμε πάνω από το μέσο ποσοστό για την ε, ε, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι υπερβολικά ακραίο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και ο κύριος Κόφωτ παρακαλώ. Κόφωτ, ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την προαναγγελία ότι θα συνεχιστούν οι συζητήσει το Σεπτέμβριο. Επικοδομητικό Ευχαριστώ κύριε Κανιέτε για μια πολύ καλή παρουσίαση. Θα είμαι πολύ σύντομο. Πρώτα στην απάντηση προς ε, τον κύριο Κάρινς είπατε είναι σημαντικό, αν σας κατάλαβα σωστά, για τον ρόλο του ΕΣΑΡ. Θέλουμε να ενισχυθεί αυτός ο θετικός ρόλος και για το θέμα των τεχνητών αυτών ε, ε, καταστάσεων που δημιουργούνται θα δώσετε εντολή στο ΑΕΣΑΡ να αντιμετωπίσει αυτές τις τεχνητές στενοπούς διότι θα πρέπει να σχεδιαστεί αυτό για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Πρώτο. Δεύτερο, θα ήθελα να πω, ίσως από πλευράς προσέγγισης να το λάβουμε περισσότερο υπόψη. Θα συνεχιστούν σε σχέση με τα πιστοποιητικά ή ε, κάποια ελεύθερα πιστοποιητικά και λέτε ότι ταυτόχρονα θέλουμε να είμαστε πρωτοπόροι στα ΑΠΕ. Πώς θα μπορέσει να γίνει το ένα με το άλλο και να συνδυαστούν. Είναι κάπως αντιφατικά το ένα με το άλλο. Και τέλος, για την οδηγία για την ετικετοποίηση δεν, είναι, δεν δημιουργεί κάποια σύγχυση ότι για τους καταναλωτές το νέο σύστημα θα υπάρξουν ε, κάποιες, ε, κάποια προβλήματα ή σύγχυση όταν έχουμε ε, το α και το β που όπως προτείνεται όμως δεν θα προβλέπεται τελικά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ συνάδελφε. Ο κύριος Ρόιλ παρακαλώ. σε αντίθεση με τον Τούρμες δεν είμαι καθόλου ενθουσιασμένος με τις προτάσεις σας. Πρώτον όσον αφορά την ιστορία με την ετικετοποίηση. Σε κάποιες συσκευές ε, που υπάρχει αναγκαιότητα να υπάρχει σαφήνεια για τους καταναλωτές το τι γίνεται, μπορεί να γίνει αυτό χωρίς αναδιατύπωση της οδηγίας. Ούτε χρειάζεται κάποια ψηφιοποίηση, ούτε κάποια μητρώα, απλά και μόνο να μπορέσουμε με το συν-συν να δημιουργήσουμε μια νέα ε, κατάσταση για αυτές τις συσκευές. Γιατί να κάνουμε ένα ε, ευρύτερο πλαίσιο για όλα αυτά. Δεύτερον, στις εκπομπές ρήπων θα πρέπει η δική μας ε, Επιτροπή να συμμετέχει στη, ε, όπως πρέπει σε αυτό το θέμα και να μην μας εκπροσωπεί η Επιτροπή ε, Περιβάλλοντος ή να, μας υποκαθιστά. Δεν πρέπει να ε, υπονομευτεί η βιομηχανία και οι επιχειρήσεις. Πρέπει να σταθμιστούν όλα αυτά προσεκτικά ποιες είναι οι επιπτώσεις τους στις επιχειρήσεις. Το κόστος και η επιβάρυνση μονοβαρός επιβαρύνουν τις βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις. Για τα πιστοποιητικά όλα επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι ευφυές όταν ζητούμε να υπάρξει ευφυής ανάπτυξη και όταν έχουμε και τα προβλήματα της Ελλάδας. Δεν νομίζω να ταιριάζουν όλα αυτά. Thank you very much, Ευχαριστώ συνάδελφε. Και επόμενος. Μαραγκάλ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ακούσαμε πολύ θετικά τις εκφράσεις που χρησιμοποιήσατε αναγνώρισης και για το μέλλον και όσον αφορά την ανάπτυξη στα ΑΠΕ, ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στα ε, ενεργειακά μείγματα, μίξ και ταυτόχρονα εκφράσεις προστασία λέει για την αυτοκατανάλωση γύρω από αυτά τα θέματα έτσι τοποθετηθήκατε. Άμεσα ερωτώ πώς ε, αξιολογείτε την γραμμή δράσης της κυβέρνησης που γνωρίζετε καλύτερα της Ισπανικής κυβέρνησης όσον αφορά την πρόβλεψη νέων ρυθμίσεων με σοβαρές κυρώσεις ή ε, ποινές που θα συνεπάγεται η δημιουργία αυτών των προτάσεων σε σχέση με δίκτυα μη φυστάμενα. Και όλα αυτά από πλευράς της ίδιας κυβέρνησης που ζητεί να υπάρξουν κυρώσεις και ποινές αναδρομικές σε σχέση με τα όσα έπρεπε να είχαν γίνει για τα ΑΠΕ. Εδώ υπάρχει μια προφανής ε, αντίφαση και από πλευράς της ε, κυβέρνησης της Ισπανίας ε, δεν ζητείτε μια εγκατάλειψη αυτού του κριτηρίου και μια αλλαγή πολιτικής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ συνάδελφε. Η κυρία Ντεκαστήγιο, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε για την παρουσίαση των προτάσεων. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τη συζητήσουμε το Σεπτέμβριο. Παρ' όλα αυτά θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Φυσικά υποστηρίζω τη γραμμή που <clears throat> παρουσίασε ο συνάδελφος Ρόιλ για την επαναβιομηχάνηση και τις επιπτώσεις που πρέπει να έχει μια ανάπτυξη και των, της, των εκπομπών ρήπων. Αλλά πρέπει να δούμε και το λιανικό, εμπόριο εδώ και να υπογραμμίσουμε την θεμελιώδη σημασία που έχει η στάση των καταναλωτών όσον αφορά την αγορά ενέργειας. Και, ε, μετά στο τέλος τέλος ε, λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία για τον καταναλωτή για να μπορέσει να δράσει και να διαμορφώσει την κατανάλωση ενέργειας από πλευράς του υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο αν δεν συμπεριληφθεί θα υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις. Η διαλειτουργικότητα είναι αυτό το στοιχείο. Η διαλειτουργικότητα είναι σημαντικό στοιχείο και εδώ πρέπει να υπάρξουν προδιαγραφές ε, για να λειτουργήσει η διαλειτουργικότητα. Θα πρέπει να υπάρξουν επιλογές για τους καταναλωτές και μέσω της διαλειτουργικότητας ε, το βασικό πρότυπο δεδομένων που θα καθορίζει τις ανάγκες των καταναλωτών θα είναι αναγκαίο να είναι φορητού χαρακτήρα, να μπορεί να μεταφερθεί, να έχουμε βασικά πρότυπα που θα καθορίζουν έτσι την στάση και ε, αντιμετώπιση του κάθε χρήστη. Και έτσι λοιπόν με αυτές τις προδιαγραφές να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Mr. Commissioner Κύριε Επίτροπε, να σας δώσουμε ένα λεπτό για να προετοιμαστείτε. Όχι, το τελευταίο ερώτημα ήταν πολύ συγκεκριμένο. Και σκεφτόμουν πώς να το απαντήσω. Θα προσπαθήσω να τα απαντήσω όλα όμως. Υπήρξε μια πρώτη παρατήρηση από την κυρία Γκρίφιν, αν δεν κάνω λάθος, για την ενεργειακή ανέχεια τα επίπεδα ενεργειακής φτώχεια στην Ευρώπη είναι τόσο ψηλά που 11% των Ευρωπαίων δεν έχουν τα χρήματα για να θερμάνουν τα σπίτια τους. Πρέπει να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Η Κομισιόν θα εξετάσει πώς μπορεί να βελτιώσει την συλλογή δεδομένων για την παρακολούθηση της ε, ενεργειακής ανέχειας και θα εξετάσουμε ελάχιστα κοινά κριτήρια για την αντιμετώπιση ε, της τροτότητας ορισμένων ε, καταναλωτών. Υπάρχουν ορισμένες υφιστάμενες ε, πρωτοβουλίες και ενέργειες. Συνεργαζόμαστε με μια ομάδα για τους ευάλωτους καταναλωτές που έχει γίνει από το Citizens Energy Forum και έχουμε ως στόχο να αναπτύξουμε λύσεις ε, για την ε, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε ό,τι φορά τους ευάλωτους καταναλωτές. Πρότασή μας είναι να υπάρξει στοχευμένη στήριξη ε, που ε, να παραέχεται κυρίως μέσω ε, κοινωνικών μέτρων και όχι προτιμησιακών χρεώσεων μπορεί να δώσει αρνητικά κίνητρα σε ό,τι αφορά την ενεργειακή απόδοση. Επίσης, ρωτήσατε κατά πόσο, τι γίνεται, ποια είναι η θέση μας για την, για την αυτόνομη κατανάλωση. Εμείς στηρίζουμε αυτό το στόχο, έχουμε εντοπίσει βέβαιες πρακτικές σε ένα staff working document που συνοδεύει την ανακοίνωσή μας και αυτό το έγγραφο δείχνει πώς μπορεί να ενθαρρυνθεί αυτή, αυτού του είδους η κατανάλωση. Είναι ένα πρώτο βήμα. θέλουμε να ακούσουμε και τις απόψεις των ενδιαφερομένων για να δούμε αν θα το θίξουμε αυτό το ζήτημα σε μελλοντική νομοθεσία για το self-consumption. Θα γίνει διαβούλευση και μάλλον και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα το συμπεριλάβει και στην νομοθεσία, που μάλλον θα έρθει ε, το δεύτερο εξάμενο του 16. Θα υπάρξει λοιπόν τότε νομοθεσία αυτό το ζήτημα. Ένα ερώτημα είχε θέσει ο κύριος Μαραγάλη. Για το σχέδιο ε, διατάγματος στην Ισπανία για την ε, αυτοκατανάλωση της 5ης Ιουνίου έχει ως αρχή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην τοποθετείται επί τέτοιων ε, σχεδίων προτού εγκριθούν. Όταν θα έχουν εγκριθεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλύσει τη συμβατότητα αυτών των μέτρων με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και θα ανακοινώσει στις Ισπανικές Αρχές τις παρατηρήσεις της <clears throat> αν υπάρξει κάποια ας το πω έτσι παραβίαση ή μη ευθυγράμμιση με τις ε, κοινοτικές αρχές. Και σε σχέση με την θέση της Επιτροπής ε, κάνατε μια παρέμβαση για τις νέες διατάξεις όσον αφορά την υποστήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε σχέση με την Ισπανία υλοποιεί τις υποχρεώσεις της και βρίσκεται και πάνω κατά 7% από ε, τις προβλεπόμενες επιδόσεις ε, σε σχέση δηλαδή με, την, ε, με τη στοχοθέτηση. Θα παρακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εξέλιξη για να δούμε αν, τι θα γίνει με τις επιδόσεις. Πρόκειται για μια διπλή ανάλυση αυτών των διαγραφών. Αφενός αυτή η μεταρρύθμιση που δρομολογήθηκε για να, να ελέγξουμε, να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των ελλείψεων όσον αφορά τον, τα τιμολόγια θα πρέπει σε σχέση με τα ανανεώσιμα να αναλυθεί. Αναλύει αυτή τη μεταρρύθμιση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν υπάρξει παραβίαση κάποιας ευρωπαϊκής αρχής θα αναλάβουμε τα ενδεδειγμένα μέτρα. Αλλά επιπλέον <clears throat> ειδοποίησε η Ισπανική κυβέρνηση για το νέο αυτό σύστημα υποστήριξης όσον αφορά τα ανανεώσιμα και αναλύεται αυτό μέσα στο πλαίσιο των επιδοτήσεων και των ενισχύσεων όσον αφορά τα πλαίσια ανταγωνισμού για να δούμε αν συνάδει με, την, με τις αρχές της εσωτερικής αγοράς. Δύο διαδικασίες έχουμε λοιπόν όσον αφορά τα θέματα ανταγωνισμού από πλευράς της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού και τα θέματα της Γενικής Διεύθυνσης για τα θέματα ενέργειας. Υπήρξε και ερώτηση προηγούμενα για την της ε, ε κυρίας Ευρωβουλευτού όσον αφορά τις ε, τιμές καταναλωτών και την ενημέρωση σχετικά των καταναλωτών. Είναι σαφές ότι θα πρέπει σε σχέση με την ενημέρωσή τους να είναι σε θέση να αντιδράσουν σε σχέση με τη διαμόρφωση τιμών. Και ένα δυναμικό σύστημα τιμών θα δίνει τη δυνατότητα να υποφεληθούν από αυτές τις ευκαιρίες οι καταναλωτές. Αυτό απαιτεί ένα συγκεκριμένο μικρής εμβέλειας ε, δίκτυο και μικρούς μετρητές. Όμως ε, η το τμήμα αυτό των μικρών μετρητών θα πρέπει να βρίσκεται σε αναλογία με τις προσφορές της αγοράς και οι υποδομές αυτές σε σχέση με τους μετρητές πρέπει να διασφαλίζουν την τεχνική διαλειτουργικότητα και η κυρία Πιλάντερ Καστίγιο το ανέφερε αυτό να υπάρχει πρόσβαση σε σχέση με στοιχεία των καταναλωτών να μπορούν έτσι διαλειτουργικά να αντιμετωπιστούν. Έχουμε δουλειά να κάνουμε εδώ λοιπόν και αν τα ε, ε, όργανα τυποποίησης ε, και εναρμονισμού πρέπει να αντιμετωπίσουν κάποια θέματα για τα small grids, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθήσει αυτές τις προδιαγραφές εκ του σύνεγγης και θα αναλύσει αν οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές για αυτά τα δίκτυα grids και για τους μικρούς μετρητές συμμορφώνονται οι χρήστες με αυτά για να υπάρχει διαλειτουργικότητα. Διότι οι προδιαγραφές και η διαλειτουργικότητα είναι σημαντικά στοιχεία και για, την, ε, ε, για τις επαφές ε, και συνεννόηση ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να λειτουργήσουν όλα αυτά σωστά. Υπάρχει ένα ολόκληρο πλέγμα δυνατοτήτων εδώ και πρέπει να το παρακολουθήσουμε. Έγινε λόγος μακροπρόθεσμα για τον, από τον κ. Μάρτιν Πιστεύουμε στη μακροπρόθεσμη αυτή προσέγγιση και στην διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους αυτό που κάναμε ήταν θεσπίσαμε, καθορίσαμε ένα ερωτηματολόγιο με 20 ερωτήσεις ερωτήσεις προς τους χρήστες. Είπαμε, μακροπρόθεσμα τέτοιες συμβάσεις ε, χρειάζονται ώστε να διασφαλιστούν οι επενδύσεις Ποια προσκόμματα είναι εκείνα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Υπάρχει ρόλος για το δημόσιο τομέα ώστε να μπορέσουν οι αγορές να συμμετάσχουν σε τέτοιου είδους μακροχρόνιες συμβάσεις. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν το θέμα, μένουμε τις απαντήσεις ε, των χρηστών και των εμπλεκόμενων και έτσι θα δράσουμε. Υπήρξε επίσης και το ερώτημα των ε, ε, μέτρων που διασυνοριακά πρέπει να ληφθούν και θα σας δώσω την ίδια απάντηση που λαμβάνουμε πάντα σε σχέση με την αντιμετώπιση των προβλημάτων και στην παρέμβαση του κυρίου Μάρτιν. Υπάρχουν εδώ κάποια ζητήματα, η εφαρμογή είναι δύσκολη υπόθεση για, την, ε, ε, για τα εισαγόμενα και την ανταπόκρισή τους ε, στις προδιαγραφές και πρέπει εδώ οι αντιδράσεις των εμπορικών εταίρων να ληφθούν υπόψη. Έτσι βράχει πρόθεσμα ο καλύτερος τρόπος είναι να υπάρχουν ποσά τα οποία θα μπορούν να υπολογιστούν σε σχέση με αυτές τις βιομηχανίες ώστε να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις ε, της Συμφωνίας για την Προστασία του Κλίματος έναντι άλλων που θα πρέπει και αυτοί να συμμορφώνονται με αυτές ε, και σε σχέση με μια αγορά που λέει δεν λειτουργεί αγορά ε, άνθρακα Πρέπει να δούμε εδώ την μείωση των εφομών ρήπων που ε, δημιουργεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Αυτή τη μεταρρύθμιση προσπαθούμε σε αυτό το πλαίσιο να την αντιμετωπίσουμε. Είπε ο κύριος Κόφωτ ότι πρέπει τα προβλήματα να αντιμετωπιστούν ως Ευρωπαίοι ρυθμιστές πρέπει να έχουμε νέο δυναμικό για να αντιμετωπίσουμε την περιφερειακή συνεργασία και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις στενοπούς όσον αφορά τις ροές ενεργειακών προϊόντων. Θα πρέπει να υπάρχουν οι πληροφορίες και να δούμε στη μελλοντική νομοθεσία κατά πόσον θα, θα κάνουμε προτάσεις για να αντιμετωπιστούν τα θέματα μέσω περιφερειακής συνεργασίας και ε, περιφερειακών ή τοπικών στενοπών. Και για την άρση ή την κατάργηση της μεγάλης κατηγορίας πρέπει να πούμε ότι τώρα έχουμε ένα περίπλοκο σύστημα με α συν, α συν συν και α 3 συν αντί του α β γ δ και έτσι λοιπόν θα εξαπλουστευτεί το σύστημα και θα έχουμε συσκευές που με αυτή την ετικετοποίηση θα γνωρίζει κανείς ότι παίρνει το καλύτερο προϊόν που είναι διαθέσιμο. Όταν παίρνει σήμερα για παράδειγμα κάποιος ένα α συν ή α συν συν μπορεί να έχει διαφορά από το πιο προηγμένο προϊόν. Ο κύριος Ρόι λέει ότι σωστά ότι η κοινοβουλευτική σας επιτροπή πρέπει να εμπλέκεται στην ε, εκπόνηση αυτών των προτάσεων. Σωστό αυτό. Πρέπει εδώ αφοράται και η ευρωπαϊκή βιομηχανία που ε, εμπλέκεται σε αυτή την, από αυτή την νομοθεσία εταιρείε που έχουν την έδρα του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα υποστούν τι επιπτώσει αυτών των μέτρων. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα αντιμετωπιστούν τα θέματα διαρροή άνθρακα. Η δική σα επιτροπή είναι η πιο ενδεδειγμένη και θα συμμετέχει. Ο κύριο Ρόιλ θεωρεί ότι είναι πολύ περίπλοκο το θέμα τη οδηγία για, ε, για την ετικετοποίηση. Θέλει να πλουστευτούν τα πράγματα. Να υπάρξει ένα κανονισμό καλύτερα και όχι οδηγία που θα εφαρμόζεται από τα κράτη-μέλη. Πιστεύουμε ότι εδώ για το σκοπό που θέλουμε πρέπει να επιλέξουμε το πιο σωστό μέσο. Θα αναμείνουμε την πρόταση του Κοινοβουλίου να διατυπωθεί και θα δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε και εμείς τη δική μας πρόταση. Ο στόχος μας όμως είναι να πλουστεύσουμε και να περάσει ένα σαφές μήνυμα προς τους πολίτες και να είναι εύκολο στην εποπτεία να γίνεται ο έλεγχος, να μην υπάρχουν παραβιάσεις ε, των διατάξεων για την ετικετοποίηση, γιατί αυτή τη στιγμή είναι πολύ εύκολο να παραπλανήσει κανείς ή να εξαπατήσει λέγοντας ότι κάποιες συσκευές για παράδειγμα έχουν τις βέλτιστες επιδόσεις. Για παράδειγμα, όταν θα υπάρξει η νέα βάση θα μπορεί αμέσω κανεί να ελέγξει. Απλουστεύουμε και είναι πιο εύκολο ο έλεγχο. Φυσικά βέβαια θα, μπορούν, θα μπορεί αρχικά να υπάρχει κάποια αρχική σύγχυση. Όμω, ανάλογα με τα κράτη-μέλη που θα έχουν ε, καλύτερε επιδόσει, όπω η Αυστραλία σε αυτά, είδαμε ότι ήταν πολύ μικρή η σύγχυση και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών δεν απολέστηκε, δεν χάθηκε. Μπόρεσαν οι καταναλωτές μετά την αλλαγή συστήματος και ε, νομοθετικής ρύθμισης να προσαρμοστούν εποφελώς. Και υπήρξε και μια ερώτηση αν θα υπάρξει ε, κάποια συσκότηση ή δεν θα λειτουργήσει το ηλεκτρικό δίκτυο σε σχέση με την παραγωγή δυναμικού ε, ως θέμα αρχής πρέπει να πω ότι για τις αγορές θα πρέπει να είναι σε θέση να παράξουν το αναγκαίο δυναμικό χωρίς ε, να υπάρχει εδώ η ανάγκη να ε, λειτουργήσουν γεννήτρες και τα λοιπά. Όμως ε, με την, τον σχεδιασμό αγορών προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια πιο αποτελεσματική αγορά ώστε να αποφευθούν και μηχανισμοί στρέβλωσης της ελεύθερης ροής ηλεκτρικού ρεύματος και να μπορέσουμε να είμαστε το δυνατό πιο αποτελεσματικοί και στο περιφερειακό και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα δούμε πόσο μακριά και ποιες θα μπορεί να είναι οι επιδόσεις μας και πόσο μακριά θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ε, υπάρχουν συζητήσεις ε, μακρότατες και χρονοβόρες, έχουμε προτάσεις ε, στο τραπέζι και όλα αυτά χάρη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε πρόκειται για το νέο σχήμα και την αγορά, το νέο σχεδιασμό για την ηλεκτρική ενέργεια, για τις ηλεκτρικές συσκευές πάλι της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας ή με το σύστημα εκπομπής ρήπων που και αυτό αφορά τις Ευρωπαϊκές Βιομηχανίες. Προσπάθησα να είμαι το δυνατό περιεκτικότερος πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Είναι προφανέ ότι δεν επαρκεί ο χρόνο για μια τέτοια συζήτηση στην Επιτροπή μα. Θα θέλαμε να έχουμε περισσότερο χρόνο ομιλία και για τα μέλη μα όπως μου το ζητήσατε κι εσείς και το κατανοώ. 21-22 Σεπτεμβρίου, συνάδελφοι, ας είμαστε έτοιμοι τότε να εξετάσουμε αυτό το θέμα ακόμα περισσότερο και σε μεγαλύτερο βάθος. Γιατί είναι τρεις προτάσεις που έχουν τεθεί επιτάπητος και είμαστε υπεύθυνοι και αρμόδιοι για όλες ως Επιτροπή Ήτρε. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να καλέσουμε τον κύριο Επίτροπο για τις 21 και 22 Σεπτεμβρίου. Θα δούμε τώρα πότε βολεύει και τον Επίτροπο να έρθει. Ακριβώς μετά τις διακοπές λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Επίτροπο, για την παρουσία σας εδώ σήμερα, για την πολύ καλή αυτή συζήτηση. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους που μείνατε εδώ για μια μισή ώρα. Και τώρα ε, να δω με τους ε, συντονιστές αν μπορούμε να κλείσουμε ε, μέσα σε μισή ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ τους υπόλοιπους. Τα λέμε αύριο στις 9 το πρωί. Start as quick possible as possible. Ας ξεκινήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα την ε, συνεδρία των συντονιστών συνάδελφοι.